Συνάδελφοι, άρχεται η συνεδρίαση. Πρώτα απ' όλα, να καλωσορίσω τον πρώην συνάδελφο, τον κύριο Στόκμαν και πάντα είναι ευχάριστο να βλέπουμε εδώ πέρα πρώην συναδέλφους. Καλώς ήρθες, Ούλη έγκριση του σχεδίου ημερήσια διάταξης που έχετε μπροστά σας. Υποθέτω πώς εγκρίνεται. Εάν ναι, περνάμε στα πρακτικά τη συνεδρίασης 1η ε, και 2 η Δεκεμβρίου 2009. Εγκρίνονται και αυτά. Ωραία, ευχαριστώ. Να υπενθυμίσω στους συναδέλφους ότι Μεταδεδόμαστε και στο διαδίκτυο και να υπενθυμίσω πως ε, την Τετάρτη έχουμε αλλαγή αίθουσας θα στο το πω και όταν τελειώσουμε θα πάμε στην 5G3 επόμενο σημείο στη μερίσια διάταξη ανταλλαγή απόψεων με τον κύριο Μπαγκέ ο οποίος ασκεί καθήκοντα διευθυντή για την εσωτερική ναυσιπλοεία. Πού βρίσκεστε? Ωραία, σας ευχαριστώ. Έχετε τον λόγο. Uh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Καλησπέρα σας. Μου, ζητήθηκε να εκπροσωπήσω την Κομισιόν, τη Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Ενέργειας, να σας ενημερώσω για το τι κάνει η Κομισιόν για τον τομέα της εσωτερικής ναυσιπλοείας με ε, ιδιαίτερο βάρος στην οικονομική κρίση που επηρεάζει τον τομέα των μεταφορών και οπωσδήποτε τις εσωτερικές ε, θαλάσσιες ποτάμιες μεταφορές. Θα ε, μιλήσω από τα λεπτά μου επιτρέπετε και μετά θα δεχτώ ερωτήσεις από τους ε, βουλευτές. Η εσωτερική πλοία, λοιπόν αποτελεί τμήμα το οποίο χρησιμοποιείται πολύ λιγότερο από ότι οι οδικές μεταφορές και οι σιδηροδρομικές μεταφορές αλλά σε ένα φυσιολογικό έτος πάνω 500 εκατομμύρια τόνοι φορτίου μεταφέρονται στην εσωτερική ναυσιπλοεία και αυτό αντιπροσωπεύει 140 δισεκατομμύρια τόνους ένα χιλιόμετρο. Οπότε βεβαίως ε, όσον αφορά το συνολικό όγκο του φορτίου που μεταφέρεται είναι αρκετά σημαντικό. Είναι ένα 5% του φορτίου που μεταφέρεται σε Ευρωπαϊκή Ένωση. Προφανώς σε κάποιες περιοχές, γιατί δεν έχουν όλες οι περιοχές αυτό το προνόμιο. Σε κάποια κράτη-μέλη λοιπόν μπορεί το ποσοστό της εσωτερικής ναυσιπλοείας να είναι πολύ πιο σημαντικό και αυτό ισχύει ειδικά για την Ολλανδία όπου βεβαίως ε, εκεί πέρα η εσωτερική ναυσιπλοεία αντιπροσωπεύει το 40% των ε, εσωτερικών μεταφορών και απασχολούνται 30.000 άνθρωποι και συχνά είναι αυτοαπασχολούμενοι σε 7.000 εταιρείες, συχνά οικογενειακές. Οπότε η εσωτερική ναυσιπλοεία έχει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα και ειδικά όσον αφορά τις χίδιν μεταφορές με χαμηλό κόστος. Τα τελευταία 10 με 20 χρόνια βεβαίως έχει μπει σε μια νέα αγορά, αυξάνει το ποσοστό της μεταφορές εμπορευματοκιβωτίων με μια ανάπτυξη μέχρι την κρίση ετήσια κατά 20%. Τα κοντέινερ δηλαδή εκτός των χίδιν μεταφορών έχουν μια συνεχή αύξηση. Όπως ξέρετε η εσωτερική ναυσιπλοεία δεν είναι μόνο φτηνή αλλά και ειδικά έχει χαμηλή κατανάλωση ενέργειας και εκπομπές οπότε είπα γύρω στο 5% των μεταφορέν και είναι λιγότερο από το 100 των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα των μεταφορών, οπότε βλέπετε πως η ενεργειακή αποτελεσματικότητα είναι πολύ υψηλή και τέλος πρέπει να σημειώσουμε πως ε, υπάρχει αρκετό δυναμικό ανεκμετάλλευτο ακόμα και εκεί όπου υπάρχει συμφόρηση στον Δούναβη, παραδείγματο χάρη στον Ρήνο ή στον Ροδανό δεν υπάρχει πρόβλημα όσον αφορά την ε, δυναμικότητα του ποταμού πλην ορισμένων στενοπών. Οπότε είναι ένας τρόπος ε, μεταφοράς ε, τον οποίο έχει αναγνωρίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση ως πολύ σημαντικό και αποτελεσματικό και έχουμε πει σαφώς Λευκή Βίβλο του 2001 αλλά και του 2006 πως η εσωτερική ναυσιπλογία πρέπει να στηριχθεί και είναι επιθυμητό να αυξηθεί το ποσοστό που έχει στις μεταφορές. Επίσης είχαμε πει το 2001 και το 2006 πως προφανώς για να συμβεί κάτι τέτοιο σημασία έχει και η καλύτερη ενσωμάτωση της στην όλη αλυσίδα του εφοδιασμού και βεβαίως ε, δεν θα σας ε, προξενήσει έκπληξη πως αυτή την προσέγγιση ακολουθούμε και στην αναθεώρηση της ε, πολιτικής μας και βεβαίως δεν το είχαμε αναφέρει στην ανακοίνωση του Ιουνίου αλλά είναι πίσω από την διαδικασία για το μέλλον των μεταφορών που ξεκινήσαμε το 2009 πέρα από αυτό το γενικό πλαίσιο θα γνωρίζετε πως υπάρχει μια συγκεκριμένη δράση, το πρόγραμμα Ναϊάδες, που συμπεριλαμβάνει μέτρα νομικής φύσης, στήριξης και συντονισμού όσον αφορά τις συνθήκες αγοράς, τον στόλο, τις ε, θέσεις εργασίας ε, και τις υποδομές καθώς επίσης και τις δεξιότητες. Οπότε τρέχει το πρόγραμμα μέχρι το 2013 και θα γίνει μια μεσοπρόθεσμη αναθεώρηση του προγράμματος για να αξιολογήσουμε την αποτελεσματικότητά του και δεν έχω καμία αμφιβολία πως στο μελλοντικό πλαίσιο που ανέφερα πριν ε, και για τους διευρωπαϊκούς, τα διευρωπαϊκά δικτύα θα ε, στηρίξουμε ως ε, Κομισιόν την εσωτερική πλέον. Τώρα για την ε, οικονομική κρίση και τον αντίκτυπο που είχε να πω πρώτα απ' όλα πως η κρίση αυτή χτύπησε τις μεταφορές αδιάκριτα οδικές, σιδηροδρομικές, αεροπορικές και θαλάσσιες και είχαμε μεγάλη μείωση των, του όγκου που μεταφέρονταν 20 ε, με 30% και ανάλογη μείωση των εσόδων. Και αυτό ισχύει για όλο το σύστημα μεταφορών και όλους τους τρόπους μεταφορών. Ο τομέας ιστορικής ναυσιπλοείας επίσης επλήγει ιδιαίτερα λόγω της δομής του και ειδικά επειδή πολλές από αυτές τις επιχειρήσεις είναι πολύ μικρές και ευαίσθητες, ευπαθείς, αλλά και γιατί ε, σχετίζεται με την ε, παραγωγή που επίσης επλήγει. Οπότε αυτός ο συγκεκριμένος τομέας ε, έχει νιώσει τα αποτελέσματα της ε, κρίσης και ήδη υπάρχει δυσκολία όσον αφορά την πρόσβαση σε πίστοση ε, ως αποτέλεσμα και της τραπεζικής κρίσης. Οπότε τώρα πολλές εταιρείε <coughs> σε πολλά κράτη που έχουν εσωτερική έχουν προβλήματα ρευστότητας και σύμφωνα με τις τράπεζες μέχρι και 60% των εταιριών στην Ολλανδία αντιμετωπίζουν ήδη προβλήματα με τις πληρωμές τους. Και σύμφωνα με τις ε, τράπεζες η κατάσταση αναμένεται να χειροτρέψει και το ποσοστό αυτό να ανέβει. Οπότε υπ' αυτές τις συνθήκες ε, τα κράτη-μέλη πρώτα απ' όλα επεμβαίνουν και αναλαμβάνουν δράση και αυτό έγινε με όλα τα μέσα μεταφοράς μέσω των προγραμμάτων ανάκαμψης των κρατών μελών που όπως ξέρετε συντονίστηκαν σε ευρωπαϊκό επίπεδο στο Ευρωπαϊκό Σχέδιο Ανάκαμψης παρόλα αυτά στη εσωτερική ναυσιπλοεία η κρίση έχει διαφορετικό αντίκτυπο ανάλογα με το κομμάτι της αγοράς και όπως ξέρετε υπάρχουν δύο διαφορετικά Ήδη έχουμε το ξηρό και το υγρό φορτίο και είναι διαφορετικός ο αντίκτυπος στα δύο αυτά κομμάτια της αγοράς επίσης υπάρχει διαφορά μεταξύ των κρατών μελών και τα κράτη-μέλη αυτά κατ' ουσίαν είναι η Ολλανδία, το Βέλγιο, η Γερμανία, η Γαλλία και η Αυστρία. Οπότε είναι μεικτή η εικόνα μεταξύ των δύο αυτών τομέων και των πέντε κρατών μελών. Τα κράτη-μέλη τα οποία επλήγησαν ε, χειρότερα όσον αφορά την εσωτερική ναυσιπλοή είναι η Ολλανδία, που είναι και το κράτος με το μεγαλύτερο ποσοστό και το μεγαλύτερο στόλο, εκεί όπου είναι σημαντικότερος επίσης ο κλάδος για τις μεταφορές. Και αυτό το οποίο κατέστησε αυτή την κρίση πιο δύσκολη στο να αντιμετωπιστεί είναι το ότι γύρω στα 160 νέα πλοία είχαν παραγγελθεί πριν την κρίση και να φυγούνται αυτή τη στιγμή και θα τεθούν σε λειτουργία το 2010 και θα προσθεθεί και νέο δυναμικό στην αγορά δίπλα στο υπάρχον που λόγω της χαμηλής ζήτησης ούτως ή άλλως η προσφορά είναι πάρα πολύ μεγάλη. Υπ' αυτές τις συνθήκες η Ολλανδική κυβέρνηση ειδοποίησε την Κομισιόν για πιθανή στρέβλωση της αγοράς και ζήτησε από την Κομισιόν να εξτάσει τα κατάλληλα μέτρα. Οπότε αυτή τη στιγμή αναλύουμε την κατάσταση μαζί με τα κράτη-μέλη. Η ακρόαση έλαβε χώρα τον Νοέμβριο για τα αποτελέσματα της κρίσης στην εσωτερική ναυσιπλοεία. Είχαμε γύρω στα 100 άτομα από ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και η Επιτροπή του Ρήνου και ε, η συνεδρίασε μετά η Επιτροπή ε, Εσωτερικής Ναυσιπλοείας των Κρατών Μελών στις 7 Ιανουαρίου. Στο συμπέρασμα κύριε Πρόεδρε. Η πλειοψηφία των κρατών μελών συμφωνεί με την άποψη πως η κρίση αυτή, αν και επηρεάζει ιδιαίτερα τον τομέα αυτών στην Ολλανδία, δεν θεωρείται διαρθρωτική κρίση, αλλά κυκλική κρίση που επηρεάζει όλα τα μέσα μεταφοράς. Οπότε σε αυτό το πλαίσιο διαρθρωτικά μέτρα όπως ε, το να παροπλιστούν πλοία ή να υπάρξει αντικατάσταση παλιών με νέα δεν ε, ε, είναι το ιδανικότερο με βάση αυτή την ανάλυση. Όμως, όσον αφορά τα μέτρα τα οποία είναι η καλύτερη απάντηση, η Επιτροπή των κρατών μελών για την ιστορική ναυσιπλοεία συνέστησε μια επιτροπή στην οποία συμμετέχει και η Επιτροπή του Ρήνου και εκπρόσωποι του κλάδου υπό την Προεδρία της Κομισιόν και τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες θα εξετάσουμε ποια μέτρα είναι κατάλληλα για να συνεισφέρουν στην ανάκαμψη του κλάδου το συντομότερο δυνατόν. Και βεβαίω, η Κομισιόν είναι στην διάθεσή σας για να ενημερώσει την Επιτροπή σας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πακέ. Θα μιλήσουν τώρα οι εκπρόσωποι των διαφόρων πολιτικών ομάδων. Πρώτα ο εκπρόσωπος του ΕΛΚΑ. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Πακέ, η ανάλυση σας για την εσωτερική πλοία είναι σωστή. Πρέπει όμως επιτέλους να δράσουμε. Τα φορτία έχουν μειωθεί κατά 20 μέχρι 30% το τελευταίο 1,5 έτος. Αυτό σημαίνει πως ε, ειδικά οι μικρές αυτές οικογενειακές επιχειρήσεις βρίσκονται σε πολύ δύσκολη κατάσταση, το αναφέρατε, πρέπει να πληρώσουν τα δανειά τους και σε αυτή την κρίση προστίθεται και ο βαρύς χειμώνας που καθιστά αδύνατη την αυσιπλοεία σε ορισμένα κομμάτια του δικτύου. Γι' αυτό ζητάμε ακριβώς αυτός ο τομέας της εσωτερικής ναυσιπλοείας ο οποίος εργάζεται αποτελεσματικά που έχει την χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας ανά χιλιόμετρο και άρα εκπομπές να υποστηριχθεί αποτελεσματικά. Αυτό σημαίνει πως τα κράτη-μέλη από κοινού με την Κομισιόν πρέπει να διαπιστώσουν πως αυτή τη στιγμή υπάρχει μία πάρα πολύ μεγάλη οικονομική διαταραχή της αγοράς, κάτι το οποίο σημαίνει πως πρέπει να λάβουμε εξαιρετικά μέτρα. Και πρέπει να σκεφτούμε και να πούμε πως υπάρχει πλέον ένα φορτίο το οποίο, ένας όγκος φορτίου το οποίο πρέπει να μεταφερθεί. Οπότε ίσως να μπορούσαμε να ορίσουμε τιμές από κοινού ε, όσον αφορά το φορτίο για να μην οδηγηθούν αυτές οι μικρές επιχειρήσεις στην καταστροφή. Κύριε Πακέ, αναφέρατε πως ε, η απόσυρση, ας την πούμε έτσι, ε, δεν θα είναι ένα αποτελεσματικό μέσο. Όταν ε, έχουν δοθεί παραγγελίες για 160 νέα πλοία τα οποία στην επόμενη σεζόν θα λειτουργήσουν κιόλα. πρέπει να σκεφτούμε μήπως έχει νόημα να δώσουμε ένα τέτοιο πρίμα απόσυρσης όπως είχε γίνει πριν από χρόνια σε εθνικό επίπεδο. Δηλαδή τα παλαιά πλοία τα οποία σημαίνουν και παραπάνω ανεκμετάλλευτο δυναμικό να φύγουν από την αγορά και να δοθούν ευκαιρίες στις μικρότερες ε, επιχειρήσεις ε, να μην ε, χρεοκοπήσουν και να υπάρχουν μόνο μεγάλους. Τρίτον, για κοινοτική δράση, ειδικά όσον αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, νομίζω αυτό μπορεί να γίνει με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να μην υπάρξει στρέβλωση του ανταγωνισμού. Αυτά νομίζω είναι τα θέματα τα οποία κράτη-μέλη και κομισιόν πρέπει να συζητήσουν και πρέπει από την ομάδα εργασίας που αναφέρατε να αναπτυχθεί ένα σχέδιο δράσης το οποίο θα εφαρμόζει αυτά τα πράγματα και αυτό γρήγορα γιατί πάρα πολλέ επιχειρήσει και στην Ολλανδία και στη Γερμανία και στη Γαλλία είναι σε τόσο δύσκολη θέση που δεν θα αντέξουν πολύ. Η Γερμανία έδωσε κάποιες ε, δυνατότητες μέσω του Ταμείου Ανοικοδόμησης που είχε γίνει για την Ανατολική Γερμανία να δοστούν κάποιες πιστώσεις γέφυρες για να τους δοθεί μια κάποια ρευστότητα και νέες επενδύσεις. Γι' αυτό σας παρακαλώ να συζητήσετε εντατικά Κομισιόν και κράτη-μέλη τη δύσκολη κατάσταση στην εσωτερική συμπλέει. Ευχαριστώ κύριε Κιούν. Ο κύριος Αλχαντραουή για τους σοσιαλδημοκράτες. Ευχαριστώ. Έχουμε αυτή τη στιγμή μία κρίση βραχυπρόθεσμη. Βεβαίως ε, έχουμε ως γνωστόν το θετικό ρόλο μπορεί να παίξει όσον αφορά την κλιματική πρόκληση η εσωτερική ναυσιπλοεία και η σημερινή κλίση νομίζω δυστυχώς παρουσιάζει τον κίνδυνο ο τομέας αυτός να βρεθεί με κάποιο μειονέκτημα και να χάσει ποσοστό της αγοράς, κάτι το οποίο βεβαίως ε, θα διακινδυνεύσει τους μακροπρόθεσμους ε, στόχους μας. Σας παραπέμπω εδώ πέρα στο γεγονός πως μπορεί να αντιπροσωπεύει μόνο 5% ο τομέας αυτός ε, των ευρωπαϊκών μεταφορών αλλά όπως είπε και ο Κορπός της είναι μόνο 1% των εκπομπών. Δηλαδή αντιλαμβάνεστε ότι είναι 5 φορές πιο αποτελεσματικός όσον αφορά τη χρήση ενέργειας. Οπότε συμφωνώ με αυτό το οποίο είπε ο κύριος Κούν. Πρέπει πράγματι πάρα πολύ γρήγορα να δούμε Το είπατε κι εσείς ε, κύριε Πακέ πως είναι πολλές ε, μικρές ε, επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται εκεί έχουν ένα πλοίο δηλαδή κάθε μία και ε, έχουν μία μείωση 20-30-50% του, του τζίρου και βεβαίως ε, υπάρχει εδώ και αρκετό καιρό αυτή η κρίση και πράγματι υπάρχει η σχετική επιτροπή της Κομισιόν και η ομάδα εργασίας αλλά ο χρόνος πιέζει και εσείς ως Κομισιόν πρέπει να αναλάβετε την πρωτοβουλία λέτε πώς θα δούμε ποια μέτρα είναι τα ενδεδειγμένα. Ε, εμείς Θέλουμε να ακούσουμε ποια μέτρα προτείνετε εσείς στην ομάδα εργασίας για να μπορέσουμε να βγούμε από την κρίση και να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους να ξεπεράσουν την ε, κατάσταση στην οποία βρίσκονται και να ε, οδηγηθούν επιτέλους σε καλύτερους καιρούς και να μπορέσουν να δουν και κάποια ανάπτυξη. Συγκεκριμένα λοιπόν, τι σκοπεύετε να προτείνετε, γιατί λέτε πως δεν θέλετε να υποστηρίξετε την απόσυρση γιατί δεν έχουμε ε, διαρθρωτική κρίση. Τώρα ωραία το σημαίνουμε, αλλά τι προτείνετε. Δεν αμφιβάλλετε πως είναι κρίση, πως έχουν πρόβλημα οι άνθρωποι. Οπότε θέλουμε μια απάντηση. Για... Αν νομίζω αυτό θα μας βοηθήσει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Χάνες Πλασάρτ για την Άλτε. Η συντονίτριά μας, πρώτα και μετά εγώ. genau, so war das Ναι, ναι, έτσι ακριβώς. Ευχαριστώ. Νομίζω κατέστη σαφέ πω ε, ειδικά όσον αφορά την εσωτερική ναυσιπλοεία πρέπει να σκεφτούμε ακόμα πάρα πολλά πράγματα. Δεν θα το συζητήσουμε μόνο σήμερα αυτό φέτο, αλλά θα μα απασχολεί όλο και συχνότερα πάντα συζητάμε ότι πρέπει να δούμε τρόπους μεταφοράς φιλικούς προς το περιβάλλον και όλοι γνωρίζουμε πως η ναυσιπλοεία ανήκει σε αυτούς και ακριβώς όσον αφορά την εσωτερική ναυσιπλοεία ε, που συνδέει τα μεγάλα λιμάνια με την ενδοχώρα έχουμε μεγάλο δυναμικό το οποίο δεν έχει χρησιμοποιηθεί για τους χύψη λόγους. Γι' αυτό πρέπει να το δούμε λίγο πιο ζεστά το θέμα και αναμένουμε πράγματι επικοδομητικές προτάσεις από την Κομισιόν, όχι μόνο τώρα το τι θα γίνει με την κρίση αυτή που έπληξε όλα τα μέσα μεταφοράς και την ε, εσωτερική ναυσιπλοεία, αλλά να δούμε πώς ε, θα προχωρήσουμε όσον αφορά και τις ε, μεταφορές με πολλαπλά μέσα μεταφορών γιατί είναι και οικονομικός και οικολογικός τρόπος μεταφοράς, οπότε αναμένω και εγώ προτάσεις για τις οποίες ε, σας συνεργούμε. Σας ευχαριστώ. Η πράσινη, κύριο Σκράμερ. Δεν έχουμε κρίση μόνο στις μεταφορές έχουμε οικονομική και χρηματοοικονομική κρίση που χτυπάει τους πάντες. Π.χ. στη Γερμανία με την απόσυρση για τα αυτοκίνητα βεβαίως βραχυπρόθεσμα βοηθήσαμε την αυτοκίνητοβιομηχανία αλλά αυτό επέδρασε και σε άλλους. Γιατί βεβαίως ο δημόσιος πλούτος δεν ε, πολλαπλασιάζεται. Π.χ. μια οικογένεια η οποία ήθελε να αγοράσει μια νέα κουζίνα και ένα νέο αμάξι σε 3-4 χρόνια, αγόρασε τώρα αμάξι γιατί ήταν φτηνό με την απόσυρση, αλλά δεν αγόρασε την κουζίνα. Οπότε, αντιλαμβάνεστε και αυτό ισχύει για πολλούς άλλους κλάδους. Οπότε πρέπει να δούμε ακριβώ συνολικά τον τομέα των μεταφορών, ακριβώ γιατί ήταν πολύ φτηνέ οι μεταφορέ και όπως αναφέρθηκε και από το παράδειγμα από τη Μεγάλη Βρετανία τα 5 εκατομμύρια τόνων που είναι η ποσόστοση εξαγωγών και είναι ακριβώς και η ποσόστοση εξαγωγών. Μπορεί να καταργηθεί αυτό και να μην προσέξει κανεί τη διαφορά. Δηλαδή πηγαίνει και έρχεται το κρέας χωρίς νόημα. Οπότε η εσωτερική ε, ναυσιπλοεία είναι ένα λογικό μέσα εάν προσαρμοστούν τα πλοία στους ποταμούς και τηρήσουν τις οικολογικές προδιαγραφές έχουμε εδώ πέρα άδικο ανταγωνισμό υπέρ της εσωτερικής ναυσιπλοείας γιατί δεν ε, πληρώνει ούτε διόδια, ούτε ε, φόρο στα καύσιμα. Σε αντίθεση π.χ. με τους σιδηρόδρομους. Και μας είπατε 5%. Ποια είναι η εξέλιξη τα τελευταία 20 χρόνια. Νομίζω στη Γερμανία έχουμε μείωση κατά 50% τα τελευταία 20 χρόνια για να φτάσουμε στο 5%. Αυτό συμβαίνει γενικά στην Ευρώπη. Ποια είναι τα συμπέρασματα που βγάζετε. Αν υπάρχει μια δυναμία γιατί είναι μεγάλο το δίκτυο και βεβαίως είναι πάρα πολύ μεγάλη η εξάρτηση από τους ε, ποταμούς. Γνωρίζω π.χ. στον Έλβα 200 χρόνια δεν μπορεί να... 200 ε, μέρες το χρόνο δεν, μπορεί, δεν είναι πλεύσιμο ο ποταμό γιατί είτε είναι πολύ ψηλά τα νερά, είτε είναι πολύ χαμηλά τα νερά, είτε έχει παγώσει ο ποταμός. Οπότε, εντάξει, είναι χαμηλές ε, οι εκπομπές, ε, αλλά εντάξει, γνωρίζουμε τι γίνεται με την αυσιπλοεία στους ωκεανούς, που είναι πάρα πολύ κακή για το κλίμα, σκοτώνουν το κλίμα κατ' ουσίαν και είναι σκουπίδια χωρίς καν φίλτρο. Και αν συγκρίνουμε βεβαίω το τι γίνεται με την αυτοκινητοβιομηχανία και το ποιε είναι οι τεχνικέ δυνατότητε, ε, πρέπει να, να τα συγκρίνουμε. Νομίζω πω βεβαίω εδώ πέρα η κρίση αφορά συγκεκριμένα και περισσότερο την Ολλανδία. Θέλω συγκεκριμένα νούμερα. Να σου πω ότι γίνεται στη Γερμανία. 80% της εσωτερικής ναυσιπλογίας είναι στο Ρήνο. Ε, σαφές, μεγάλο ποτάμι, φαρδί ποτάμι, βαθύ ποτάμι ανεξαρτήτως ε, της, ε, δεν έχει πρόβλημα δηλαδή με την άνοδο της στάθμης και έχει πρόσβαση και στη Βαλτική και στον Ατλαντικό. Αλλά από όσο ξέρω και στην Ευρώπη 80% της ευρωπαϊκής εσωτερικής ναυσιπλοείας γίνεται στον Ρήνο. Τα λεφτά πάνε αλλού όμως. Και ονειρευόμαστε πώς θα μπουν ε, τα μεγάλα πλοία να πλέψουν στα ποτάμια και τι κάνουμε, βλάπτουμε τι μικρέ επιχειρήσει χωρί να ε, έχουμε πραγματικό αποτέλεσμα από την άλλη μεριά. Και βλάπτουμε μικρέ επιχειρήσει που έχουν μόνο ένα, ένα πλοίο στη διάθεσή του. Και αν συμβεί κάτι τέτοιο βεβαίω και υπάρξει πάρα πολύ μεγάλο πλοίο, θα πάρει αυτό όλο το φορτίο και οι μικροί θα εξαφανιστούν. Σε αυτό θα ήθελα λοιπόν μία απάντηση και Βεβαίω πρέπει να κάνουμε τη σύνδεση εδώ πέρα που αναφέρατε, δηλαδή να υπάρξει μια σύνδεση και εκεί που θα πάνε τα πλοία και με τους σιδηρόδρομους και με όλα τα υπόλοιπα και εδώ πέρα να ενδιαφέρει εδώ πέρα να δούμε τι θα γίνει με την κρίση γιατί λέμε λέμε αλλά συγκεκριμένες προτάσεις πώς θα βγούμε από την κρίση δεδομένου του ότι η εσωτερική ναυσιπλοεία μειώθηκε τα τελευταία χρόνια και πρώτης κρίση. Uh, Ευχαριστώ. Ο κύριος Βαντάλ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, το ζήτημα είναι βεβαίως το είδος της κρίσης, αναφέρθηκε από την Κομισιόν, εάν είναι διαρθρωτική ή συγκυριακή. Δεν είναι σωστή αυτή η ερώτηση, γιατί κάθε κρίση που πλήττει την εσωτερική ναυσιπλοεία είναι εξορισμού διαρθρωτική. Γιατί η εσωτερική ναυσιπλοεία ε, αντιμετωπίζει ένα ζήτημα με τον, ε, με τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της και τι εννοώ εδώ πέρα. Ένα πλοίο πλέει επί 50 χρόνια, πολύ περισσότερο από τη ζωή ενός ε, φορτηγού και ε, στην Ολλανδία στη δεκαετία του 90 είχαμε ακριβώς αυτό το μακροπρόσωπο προγραμματισμό και την απόσυρση των πλοίων λοιπά που είπαμε, ακριβώς λόγω του ιδιαίτερου χαρακτήρα. Και τώρα έχουμε φτάσει σε ένα σημείο καμπής. Επιπλέον, ο κανονισμός αυτός χρηματοδοτήθηκε από τον ίδιο τον ε, κλάδο, γύρω στα 30 εκατομμύρια ευρώ είχαν μπει στο ταμείο αυτό και ποια είναι τώρα η κατάσταση. Η Ολλανδική κυβέρνηση με τη στήριξη αυτών των επιχειρήσεων έγραψε μία επιστολή προς την Κομισιόν και είπε πως είναι τόσο σοβαρή η κρίση και τόσο πολύ χρειάζεται στήριξη της αγοράς έτσι ώστε τα δύο αυτά μέσα τα οποία έχουμε στην διάθεσή μας τη στήριξη, δηλαδή την απόσυρση και τον κανονισμό ε, θα πρέπει να τα χρησιμοποιήσουμε έτσι ώστε να βοηθήσουμε και τις επιχειρήσεις μακροπρόθεσμα να είναι βιώσιμες, αλλά τι βλέπουμε. Έχει μειωθεί πάρα πολύ και το φορτίο το οποίο πρέπει να μεταφερθεί και άρα και οι τιμές. Και βεβαίως ε, εδώ πέρα είναι ένα τομέα στον οποίο έχει η Κομισιόν το δικαίωμα τη πρωτοβουλία, αλλά τα, η πλειοψηφία των κρατών μελών σα ζητάει να λάβετε κάποια μέτρα. Οπότε η πρώτη παρατήρηση ήταν αυτή πως η κρίση είναι εξορισμού διαρθρωτική όταν μιλάμε για την ιστορική ναυσιπλοεία και δεύτερον έχει και μία δική τη ευθύνη η Κομισιόν έτσι εντός, τριών μηνών να απαντήσει στην Ολλανδική κυβέρνηση και εδώ πέρα συμφωνώ πλήρως με τον συνάδελφο Ελχαντραουή πως ε, είπε ωραία όλα αυτά τα οποία λέγεται αλλά πλέον έχει φτάσει είμαστε ίσα βάρκα ίσα νερά και δυνεύει να βυθιστεί αυτός ο κλάδος αν μου επιτρέπετε και αν δείτε τα νούμερα πραγματικά είναι ακόμη χειρότερα και το να συνεδριάζουμε και το να μιλάμε περαιτέρω δεν χρειάζεται Σα παρακαλώ λοιπόν στην Κομισιόν, χρησιμοποιήστε το δικαίωμα τη πρωτοβουλία σα, χρησιμοποιήστε τα δύο μέσα τα οποία έχετε στη διάθεσή σας, γρήγορα να βοηθήσετε την εσωτερική ναυσιπλοεία. Ε, διαρκεί τόσο καιρό αυτή η κρίση, χρεοκοπούν επιχειρήσει και μετά αντιλαμβάνεστε πως τα μέσα τη παραγωγής, δηλαδή τα πλοία εδώ πέρα εμπροκειμένα, μπαίνουν στην αγορά με καταλήγουν να είναι στην αγορά διαθέσιμα με τη μισή τιμή και η κρίση γίνεται μόνο και σοβαρότερη. Οπότε συγκεκριμένα, τι θα απαντήσετε πριν τα μέσα Φεβρουαρίου στην Ολλανδική κυβέρνηση και να δραστηριοποιηθείτε τώρα πριν χαθεί οριστικά ο κλάδος. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Φαντάλη, κύριε Βότμαν Κόλ. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για το ότι θέσατε αυτό το ζήτημα στην ημερήσια διάταξη γιατί είναι τόσο σημαντικό πως ε, πρέπει να έχουμε κατά νου αυτή τη μεγάλη κρίση και οι συνάδελφοι Ελχαντραουή και Φαντάλε ανέφεραν τη σημασία του θέματος αλλά ανέφεραν πως η ιστορική ναυσιπλοεία έχει όντως ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Και πρέπει, πρέπει να δούμε ότι αυτή τη στιγμή απειλεί και τις υγιείς επιχειρήσεις. Οπότε έχουμε πράγματι ένα διαρθρωτικό πρόβλημα, το οποίο τι σημαίνει, θα είναι τόσο εξαστετημένη η εσωτερική ναυσιπλοεία μετά την ε, κρίση, έτσι ώστε δεν θα μπορεί να παίξει αυτό τον σημαντικό ρόλο τον οποίο θέλουμε για αυτήν. Και αυτό είναι άσχημο και για την ναυσιπλοεία και για το περιβάλλον και για τις μεταφορές γενικά είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό, όπως σας είπα, να βοηθήσουμε αυτή τη στιγμή τις υγιείς επιχειρήσεις. Ε, βλέπω πως η Κομισιόν ε, ανέλαβε μία πρωτοβουλία, αλλά να τονίσω και αυτό το οποίο υπογραμμίσαμε. Εντάξει, ήμασταν ικανοποιημένοι με το πρόγραμμα δράσης Ναϊάδες, αλλά αν δούμε τώρα το τι γίνεται. Υπάρχουν πάρα πολλά μεγάλα τμήματα αυτού του προγράμματος που δεν επαρκούν και δεν έχει προχωρήσει αρκετά. Παραδείγματο, χάρη το πρόγραμμα της καινοτομία για την εσωτερική ναυσιπλοεία δεν έγινε ποτέ και είναι κρίμα πραγματικά. Και από εκεί πέρα θα γίνει τελικά και από εκεί πέρα θα προελθεί και η ενίσχυση του τομέας Και είμαι σίγουρος πως ε, η ο νέος επίτροπος, ο κύριος Κάλλας, είπε πως οπωσδήποτε θα έρθει στο Κοινοβούλιο να μας πει τι γίνεται με τις ε, ναϊάδες για να δούμε τι θα γίνει με το μέλλον της ε, ναυσιπλοείας. Αλλά εδώ πέρα βράχει πρόθεσμα πρέπει να αναλάβουμε γρήγορα μέτρα που θα έχουν αποτελέσματα γιατί η βραχυπρόθεσμη κρίση πρέπει να αντιμετωπιστεί και είμαι περίεργη και να ακούσω από πόσο γρήγορα θα μπορέσουμε να έχουμε μια συζήτηση εδώ πέρα και αποτελέσματα από αυτή την ομάδα εργασίας την οποία αναφέρατε. Ευχαριστώ. Ναι, ευχαριστώ κύριε Βαβμακόλ. Η κυρία Τίκαου. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να, ζητήσω, να ρωτήσω από την Κομισιόν εάν ξέρουν ποιος ε, ήταν ο αριθμός ε, των ε, απολύσεων στον κλάδο γιατί υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις που απέλησαν κόσμο και δεν ξέρω εάν βοηθήθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο πόσες επιχειρήσεις χρεοκόπησαν Θέλαμε, λέμε, πιο οικολογικά πλοία επίσης. Τι γίνεται με αυτό. Uh, Οπότε, θέλαμε, όπως είπαμε, πιο οικολογικά πλοία. Θέλαμε. Θέλαμε να χρησιμοποιούμε ε, αποτελεσματικά και αποδοτικά τα εσωτερικά μας ύδατα, όμως πιστεύουμε ότι θα πρέπει και η Κομισιόν να βρει μια πιο απλουστευμένη διαδικασία. Θα πρέπει να βρει τα κατάλληλα μέτρα έτσι ώστε να ε, βοηθήσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, εκτός ε, από το, τις Ναϊάδες δηλαδή και το πρόγραμμα Μάρκο Πόλο και θα πρέπει να διασφαλίσουμε επίσης και τον, τις συνδυασμένες μεταφορές. Τελευταία παρατήρηση που θα ήθελα να κάνω είναι η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το ΔΥΣΥ. Θα πρέπει, ε, πιστεύουμε, στα πλαίσια αυτής της ε, πολιτικής, η στρατηγική για την εσωτερική, εσωτερική ναυσιπλοεία να παίξει ένα σημαντικό ρόλο. Θα πρέπει να υπάρχει ένα πρόγραμμα δράσης θα πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένες ε, ενέργειες ε, με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα. Όλα αυτά τα θέματα τα οποία φύγουμε σήμερα θα πρέπει κάποια στιγμή να γίνουν πραγματικότητα. Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Τικάνη. Κυρία Χένες Πλέσιο έχει τον λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ξεκίνησε καλά την ανάλυση του εκπρόσωπος της Κομισιόν όταν είπε πως η οικονομική κρίση τους έπλεξε όλους και ειδικά την εσωτερική ναυσιπλοεία λόγω των χαρακτηριστικών του κλάδου και ανέφερε κάποια νούμερα του Σεπτεμβρίου του 2009 πράγματι Εν μεταξύ αυτό το 60% που ανέφερε έχει πάει 90% και προξενεί έκπληξη πως ε, κάνετε μια ομάδα εργασία και μετά περιμένετε και αναρωτιέμαι γιατί δεν έχει κινητοποιηθεί εδώ πέρα η Κομισιόν περισσότερο και θέλω και εγώ να ζητήσω όπως και οι άλλοι συναδελφοί μου να χρησιμοποιήσετε πλήρως όλες τις δυνατότητες που έχετε η πλειοψηφία των κρατών μελών είπε δεν είμαστε υπέρ της απόσυρσης, ε, δεν είμαστε υπέρ ε, των νέων πλοίων κτλ. Είπατε και ο ίδιος πως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι ευάλωτες και πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη ιδιαίτερο βάρος, αλλά δεν αρκεί μία ομάδα εργασίας. Δεν είναι δυνατόν για κάθε πρόβλημα να κάνετε άλλη μία ομάδα εργασίας και τελικά να μην λαμβάνετε απόφαση. Επιτέλους αναμένω πραγματικά από την Κομισιόν να καταλήξει επιτέλους σε έναν κανονισμό για την εσωτερική ναυσιπλοεία γιατί έχει μεγάλη σημασία αυτός ο τομέας και θα πρέπει να λάβει τη θέση που το αξίζει εντός της Κομισιόν και ελπίζω αυτό να γίνει με τον νέο Επίτροπο αλλά νομίζω πως δεν έχει δοθεί αρκετό βάρος και στην κοινωνία πράγματι στον ε, ρόλο της εσωτερικής ε, ναυσιπλοείας και εντάξει στην κοινωνία αλλά εντός της Κομισιόν είναι ανεπίτρεπτο γιατί πρόκειται για ένα αποτελεσματικό τρόπο μεταφορών. Ομάδα εργασία ή όχι λοιπόν, αναμένω συγκεκριμένα να προτείνει η Κομισιόν έργα τώρα, μέτρα για την κρίση. Ευχαριστώ. Κυρία Αγιάλα Σέντερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταρχάς ε, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω γιατί οργανώσατε αυτή την ε, συζήτηση και για έναν άλλον τομέα ο οποίος επλήγει πάρα πολύ σημαντικά από την κρίση ε, χαίρομαι που μιλάμε για, τα, για την εσωτερική ναυσιπλοεία. Ε, όταν συζητάμε για, την, ε, για τις μεταφορές, τις οδικές μεταφορές, κάνουμε σαν να μην υπάρχουν προβλήματα. Εγώ, πιστεύω ότι η οικονομική κρίση έχει πλήξει όλους τους τομείς, όλες, όλους τους τρόπους μεταφοράς. Η Κομισιόν θα πρέπει να ξεκαθαρίσει τα πράγματα. Πρόκειται για μια συγκυριακή κρίση η οποία θα κρατήσει ένα-δύο χρόνια κυρίως ε, πώς ε, θα μπορέσουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να έχουν την καλύτερη πρόσβαση στην χρηματοδότηση. Ή πρόκειται για ένα διαρθρωτικό πρόβλημα. Οπότε εκεί θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε με διαφορετικό τρόπο το πρόβλημα. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε περισσότερες πληροφορίες. Αυτό το οποίο μετράει βέβαια είναι να σώσουμε τις επιχειρήσεις, να διασφαλίσουμε τις θέσεις απασχόλησης των εργαζομένων. Αν υπάρχουν, υπάρχουν ε, στοιχεία που μας επιτρέπουν να δούμε τι είδους κρίση είναι, ε, θα πρέπει να, δούμε, να μας δώσει περισσότερες ε, πληροφορίες η Κομισιό για να δούμε κατά πόσον πρόκειται για μια διαρθρωτική κρίση ή όχι. Παραδείγματο χάρη εδώ έχει να κάνει και η αλλαγή του κλίματος. Η αλλαγή του κλίματος επηρεάζει τις ε, μεταφορές. Ε, θεωρούμε πάντοτε ότι η εσωτερική πλοία ε, είναι ένας καλός τρόπος, οικολογικός τρόπος μεταφορών. Όμως λόγω της αλλαγή του κλίματος μπορεί να αλλάξουν οι πλωτοί Άρα θα πρέπει να έχουμε περισσότερες πληροφορίες από πλευρά τη Κομισιόν. Επίση, αναφερθήκατε για την πρημοδότηση για τον παραπλησμό των πλοίων. Ε, δεν ξέρω αν αυτό αποτελεί μια ριζοσπαστική λύση. Εδώ μιλάμε για ένα τομέα του μέλλοντος. Μήπως ε, θα έπρεπε να δώσουμε ένα πριμ ε, το οποίο να είναι προσαρμοσμένο και στις περιβαλλοντικές απαιτήσεις μήπως ε, θα μπορούσαμε να προσαρμόσουμε τα υπάρχοντα προγράμματα ε, Πάρκο Πόλωνα, οι Άδες, ε, μήπως μπορούμε να υιοθετήσουμε νέα προγράμματα, νέες λύσεις όσο να το πιο γρήγορα για να αντιμετωπίσουμε την κρίση, έτσι ώστε ο τομέας να έχει καλύτερη και πιο εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε μια ολόκληρη γκάμα μέτρων που συνήθως του, δεν του δίδονται. Λοιπόν, μια και δεν ζητάει κανείς άλλο το λόγο, θα ήθελα να προσθέσω κι εγώ κάτι, εάν ε, γίνεται κύριε Πακέ. Εγώ ήθελα να γίνει αυτή η συζήτηση, διότι από τις αντιδράσεις ε, κάποιων συναδέλφων φαίνεται ότι ε, στον τομέα της εσωτερικής ναυσιπλοείας έχουμε σοβαρές, σοβαρά προβλήματα. Υπάρχει μια πολύ σοβαρή κρίση και το ακούσαμε από τους συναδέλφους, ήταν σαφής. Ε, όλοι είπαν ότι ήταν σωστό που είχαμε αυτή τη συζήτηση σήμερα. Όμως, όπως είπε και η κυρία Χένες Πλέσσερ, δεν είμαι σίγουρος η ομάδα εργασίας της Κομισιόν τι θα κάνει. Εγώ οφείλω να μιλήσω ότι είμαι λίγο επιφυλακτικός. Και ίσως είμαι και λίγο κοινικός τώρα και θα ήθελα να με συγχωρέσετε. Αλλά κανονικά ε, η Κομισιόν όταν αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα, έχει κάποιες, ε, κάποιες αμφιβολίες, κάποιες απορίες, λέει «Α, ας κάνουμε μία ομάδα εργασίας». Λοιπόν, δεν ξέρουμε τι να κάνουμε δηλαδή, κάνουμε μία ομάδα εργασίας. Δεν ξέρω όμως αυτή η ομάδα εργασίας τι θα κάνει, τι πρέπει να πετύχει. Γι' αυτό θα ήθελα περισσότερες πληροφορίες για το συγκεκριμένο. Γιατί για κάποιον ο οποίος δεν είναι ειδικό στην ε, εσωτερική, στην εσωτερική Εγώ το κανάλι του Μάντσεστερ ξέρω. Λοιπόν, υπάρχει μια κρίση, άκουσα, στον ε, Ρήνο. Εάν υπάρχει κρίση στο Ρήνο, στα υπόλοιπα ποτάμια μας τι γίνεται στο, στον ο, δου, Δούναβη παραδείγματος χάρη εδώ ο Ρήνος ήταν, ήταν η κόρη του, των οφθαλμών μας στην εσωτερική ναυσιπλοεία Επομένως αν εκεί υπάρχει πρόβλημα τι γίνεται στο Δούναβη ή στα άλλα ποτάμια δεν έχουμε σαφείς ενδείξεις όμως Μας είπαν κάποια στοιχεία οι Ολλανδοί, οι Βέλγοι για το τι συμβαίνει και ο κύριος Κράμερ είπε κάτι. Εμένα αυτό το οποίο ε, με εκπλήσει είναι ότι εάν οι τράπεζες, εάν οι, οι αυτοκινητοβιομηχανίες κινδυνεύουν να χρεοκοπήσουν, κανείς δεν ε, αμφισβητεί το γεγονός ότι θα πρέπει να τις βοηθήσουμε. Και δεν λέω να μην τις βοηθήσουμε, αλλά τέλος πάντων, εδώ τώρα στην εσωτερική ναυσιπλοεία ή στα άλλα μέσα μεταφορά κανείς δεν λέει πρέπει να κάνουμε κάτι συγκεκριμένο για να βοηθήσουμε αυτόν τον συγκεκριμένο τομέα οικονομικά. Τώρα δεν ξέρω πώς θα μπορούσαμε να τον, βοηθήσουμε οικονομικά. Ίσως μπορεί να είναι ο παροπλισμός των πλοίων. Δεν ξέρω πραγματικά. Όμως σήμερα δεν άκουσα τίποτα που να μου δίνει κάποιες ιδέες για το τι προτιθέμεθα να κάνουμε. Δηλαδή δεν άκουσα κάποια συγκεκριμένη ιδέα για το πώς θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε αυτόν τον τομέα ο οποίος περνάει κρίση. Και θα μπορούσαμε και μέσω τη αδράνεια βέβαια να ε, ε, πιέσουμε τον τομέα να φτάσει αν θέλετε στο, στα όρια. Αυτό όμως θα πρέπει να το αποφύγουμε. Και κάτι άλλο, γιατί θα μπορούσαν να μας κατηγορήσουν ε, σε ένα-δύο χρόνια ότι εμείς καθόμαστε και σφυρίζαμε ενώ και εγώ ήταν η Ρώμη. Επομένως θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα αυτό δίνοντάς σας το λόγο κύριε Πακέ για να απαντήσετε στα, στους συναδέλφους ε, να πω κι εγώ ότι όντως όλοι συνειδητοποιούμε ότι υπάρχει κρίση όλοι συνειδητοποιούμε ότι υπάρχει πρόβλημα και οι έξυπνοι είναι αυτοί που θα μας πούνε τι, θα, τι πρέπει να κάνουμε για να σταματήσουμε αυτή την κρίση Δηλαδή, τι πρέπει να γίνει έτσι ώστε ο τομέας της εσωτερικής να ανακάμψει. Μέχρι στιγμής ιδέες δεν άκουσα και θα ήθελα να ακούσω κάποιες τώρα ιδέες για να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε αυτόν τον τομέα να περάσει αυτές τις δύσκολες στιγμές τις οποίες αντιμετωπίσει. Και όχι να μην ε, στηριζόμαστε στον καιρό, διότι ας πούμε ε, κάποιοι υπουργοί μπορούν να ελέγξουν κάποια πράγματα ε, αλλά τον καιρό δεν μπορούν να τον ελέγξουν. Επομένως, θα πρέπει αυτός ο τομέας να βοηθηθεί να ξεπεράσει τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει. Επομένως, απευθύνω μια έκκληση. Δώστε μας κάποιο φως ελπίδας. Γιατί έτσι όπως ξεκινήσατε, στην πρώτη, η πρώτη σας παρέμβαση δεν μας έφυσε καμία, κανένα περιθώριο ελπίδας. Ελπίζω στο, εν, εντωμεταξύ να ε, βελτιωθήκατε όσο πέρασε, περνούσε και η ώρα. Ε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί βουλευτές και εγώ σας ευχαριστώ για τις ερωτήσεις σας. Πρόεδρε, δεν είμαι και τόσο σίγουρος ότι στο υπόλοιπο 5 λεπτό, 10 λεπτό που έχω στη διάθεσή μου θα μπορέσω να σας απαντήσω σε όλα αυτά που περιμένετε να σας εξηγήσω. Θα μπορέσω μόνος με κάποιες αδρές γραμμές να σας πω μια, μια διαδικασία σε σχέση με το πρόβλημα τα πράγματα οι κυβερνήσεις, οι κλάδοι, οι συναδελφοί μου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Γιατί βέβαια όλα αυτά θα προκύψουν και από τις επαφές με τον ε, Επίτροπο του οποίου είναι προτεραιότητα η ιστορική ναυσιπλοεία. Δυσκολεύομαι γιατί καταρχήν συμφωνώ με το περισσότερα από όσα είπατε. Και εγώ ανέφερα στην αρχή ότι η εσωτερική ναυσιπλοεία σαν κλάδο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ούτω ώστε να έχουμε στο σύνολο του κλάδου μεταφορών κάποιο είδου ε, πρόοδο. Νομίζουμε ότι έτσι έχουμε ένα ολοκληρωμένο σύστημα μεταφορά και έχουμε όλου του τρόπου μεταφορά που έτσι ε, θα μπορούν ε, αρμονικά να συνδυαστούν. Πρωτοβουλίε έχουμε, μέτρα έχουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εσείς έχετε προτείνει κάποια πράγματα, τα κλατιμέλη και ο στόχος είναι να μπορέσουμε να βοηθήσουμε κάποια μέτρα για να υπάρξει ένα δίκτυο εσωτερικής εμφυλίωσης που να συνδυάζεται με τους μεταφοράς και θέλουμε μέσω μακροπρόθεσμα να έχουμε ένα όραμα ώστε να μπορέσουμε η εσωτερική ναυσιπλόγια να είναι πιο πολύ πρωταγωνίστρια σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα μεταφοράς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να σα τα πω και πιο συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Βεβαίω και θεωρεί ότι είναι μια αφετηρία. Αυτό όσον αφορά το δίκτυο που θέλουμε να φτιάξουμε. Άλλωστε θα έχουν ζητηθεί και με την Επιτροπή για αυτό το δίκτυο, για αυτό το, δίκτυο το οποίο τις συνδυσμές μεταφορές θα τις έχει σε πάρα πολύ ψηλή προτεραιότητα. Θεωρείται ότι αποτελούν πύλη προς την Ένωση οι ε, λιμένες. Οπότε ήταν και θα παραμείνουν οι λιμένες εσωτερικής ναυσιπλοείας ε, και ναυσιπλοείας γενικότερα μια, ε, ένας πάρα πολύ σημαντικός παράγοντας σε αυτό το δίκτυο που θέλουμε να φτιάξουμε. Έχουμε αυτούς τους πράσινους διαδρόμους, αυτό να τους γνωρίσουμε τους αξιοποιήσουμε περισσότερο γιατί θέλουμε αυτή η αφετηρία να βοηθήσει για να έχουμε πράσινε μεταφορέ, να έχουμε πιο αποτελεσματικέ μεταφορέ, να έχουμε μια ολόκληρη αλυσίδα επιμελητία ε, για να μπορέσουμε κατά αυτόν τον τρόπο να καταφέρουμε να γίνουν αυτοί οι πράσινοι διάδρομοι οι ραχοκοκαλιές μεταφορές της Ευρώπης. Δηλαδή αυτό που το να κάνω είναι να δούμε ότι για όλους τους εμπλεκόμενους η ιστορική ναυσιπλοεία είναι ένα στόχος, μια φιλοδοξία. Γιατί έχει κάποια ενδογενή πλεονεκτήματα, όπως και έχει βέβαια ακόμα και κάποιους περιορισμού όπως ε, αναφέρθηκε. Έχουμε το θέμα των εκπομπών, αλλά πρόκειται για τρόπο μεταφοράς με πάρα πολλά θετικά και άρα μας ε, προσφέρει πάρα πολλές ευκαιρίες αποτελεσματικότητα, δεν υπάρχει διοξείδιο του άνθρακα και πέραν όλα αυτά τώρα συμφωνεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι φυσικά και υπάρχει και σε αυτό το κλάδο μια κρίση. Είναι διορθωτική, είναι κυκλική. Το θέμα είναι το τι μέτρα μπορούμε να λάβουμε σε ενωσιακό επίπεδο. Που είναι κοινωνική η κρίση, βέβαια, και τα ξέρουμε αυτά είναι ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους πέρσι οργανώθηκε η ακρόαση. Και εγώ άλλωστε προσπαθώ τώρα να σας πείσω να προχωρήσουμε προς ένα αποτελεσματικό και από κοινωνικής πολιτικής πακέτο μέτρων. Δεν έχουμε ακόμα συγκεκριμένες ημερομηνίε προβάσεις επιτροπής. πάρα πολλέ επιχειρήσει είναι οικογενειακέ, οπότε και γι' αυτό και δεν έχει φανεί ακόμα η επίπτωση στην ανεργία τη κρίση. Παρ' όλα αυτά όμω, ο κοινωνικός αντίκτυπος τη κρίση είναι πάρα πολύ σημαντικό. Άρα θα πρέπει να δούμε πώς θα έχουμε μια δέσμη μέτρα. Επίσης θα πρέπει να σα τονίσω ότι η ιστορία ψηπλοεία έχει ως η μορφή και το ότι πριν από 15 χρόνια είχε τιμές καθορισμένες, fix. Είπε πάρα πολύ αυστηρή νομοθεσία. Οπότε και υπάρχει κάποιο τρόπο μια τέτοια ανάμνηση αυτού του αυστηρού περιβάλλοντος που δεν ισχύει πια. Καθορισμός τιμών πλέον απαγορεύεται έχουμε τους, κοινωνικούς, ε, τους μάλλον κανόνες για ανταγωνισμό και κατά κάποιο τρόπο το ίδιο ισχύει και όσον αφορά ένα σύστημα το οποίο ίσχυε για χρηματοδότηση όταν έγινε η μετάβαση από την υπερβολικά ρυθμισμένη αυτή αγορά προς την σημερινή πιο απορριθμισμένη. Έχουμε προς μια σειρά μέτρων τα οποία έχουν προταθεί, τα οποία κυκλοφορούν σαν προτάσεις, ούτως ώστε να καλύψουν την κρίση και πάρα πολλές από αυτές τις προτάσεις, επομένω, ε, δεν ισχύουν πλέον διότι είτε δεν υπάρχει περιθώριο να εφαρμοστούν από την κοινωνική νομοθεσία, είτε γιατί ε, δεν συνάδουν προς αυτά τα 35 εκατομμύρια ευρώ τα οποία ε, προσφέρονται για ενισχύσεις προέβαση καλών πολλών κρατών μελών Οπότε, εάν κανείς κάτσει και κατανείμει αυτά τα κονδύλια όσον αφορά την, την απόσταση κάποιων παλιών πλοίων, θα δει ότι η κατάτμιση των ποσών φέρνει μια αποδυνάμωση του μέτρου. Και τελικά με τα χρήματα τα οποία δίδονται δεν μπορεί κανεί να κάνει απόσυρση ικανού αριθμού παλαιών σκαφών τόσο να πούμε ότι θα υπάρξει αλλαγή. Έχουμε και όλα αυτά τα μέτρα υποστήριξη. και δεν είναι θέμα δικαιώματος πρωτοβουλίας, έχουμε το θέμα το ότι πάρα πολλά ε, μέτρα προέρχονται από την αυτοκινητομηχανία, από το τραπεζικό τομέα, και έχουμε κάποια εθνικά, εθνικές προσπάθειες στήριξης. Περιμένουμε επομένω. για κάποια μέτρα εθνικά, όπως ας πούμε για τις κάτω χώρες που εμπλέκεται τόσο πολύ. Είχαμε και προτάσεις Νοέμβριο, συζητήθηκαν τον Ιανουάριο και τέτοιου είδους μέτρα στήριξης. Βέβαια ξέρουμε ότι είναι πάρα πολύ εύκολο το να πάρει κάποια κυβέρνηση. Εμείς πάντως προτιθέμεθα ανα πάση στιγμή με τους ε, Ολλανδούς να τα συζητήσουμε μόλις κατεβούν οι προτάσεις τους. Άπαξ βέβαια και είναι ε, συμβατά τα, τα, τα εθνικά μέτρα, συμβατά με το δίκαιο του ανταγωνισμού. Τόσο ώστε να πετύχουμε αυτό το οποίο θέλουμε για την πιο μακρόπνοη πολιτική μας τώρα, για κάποιο είδους μέτρα που αφορούν τις υποδομές, όσον αφορά τις πολιτικές που σήμερα ακολουθούμε, όλα αυτά τα οποία θα συζητηθούν με τον υποψήφιο επίτροπο κύριο Κάλλας, αναφέρθηκε το ποιοι είναι οι περιορισμοί που επιτάσσει η κοινωτική νομοθεσία, όμως θέλουμε να υπάρξει σχέδιο διάσωσης εθνικό. Έχουμε κοινωνικό κανονισμό, έχουμε εθνικά μέτρα, όλα αυτά θα μπορούσαν να συνδυαστούν και έτσι να έχουμε αυτή την δέσμη των σωτήρων μέτρων που θα μπορούσε να κατευθυνθεί προς κάποιο είδου ε, σύστημα πρόορες σύνταξης, προς συγχρηματοδότηση, το κοινωνικό ταμείο, όπως ξέρετε, συγχρηματοδοτεί δεν χρησιμοποιεί από μόνο του και έτσι διευκολύνει τα εθνικά προγράμματα Και επαγγελματική κατάρτιση, επαγγελματικός προσυντολισμός, όλα τα σχετικά μέτρα. Βέβαια, καλύτερη, καλύτερα τα μέτρα της ε, κατάρτισης παρά της επανακατάρτισης. Το πρόβλημα υπάρχει και θα υπάρχει πάντως έντονο και μόλις ανακαμψεί ο κλάδος από την κρίση τα επόμενα χρόνια. Ούτε θα πρέπει να δηλιάζουν. Σε σχέση και με το, το έργο που είχε αναλυφθεί όσον αφορά τα κέντρα πληροφόρηση, το πρόγραμμα Ναϊάδες, για τα της πλοήγηση, τα της ναύλωσης, της ενημέρωσης για τη μεταφορά ας πούμε των περιεκτών είπαμε ότι όλο ένα και περισσότερο αυξάνεται η διακίνηση των περιεκτών στον Ρήνο. Και επίσης χρειάζονται περισσότερη πληροφόρηση οι εμπλεκόμενοι, οι πελάτες, οι χρήστες στο σύστημα. Και αυτό και το λέμε και πιο σημαντικό. Είπαμε ότι είναι πάρα πολύ τεχνική η συζήτηση του αν έχουμε κρίση κυκλική ή διαρθωτική. Το σημαντικό είναι ότι η κρίση είναι δεδομένο. Βεβαίως, το θέμα δεδομενο Βεβαίω, το θεμα ειναι τι είδου μέτρα χρειάζονται, τι είδου αποφάσει χρειάζονται, με τι διαδικασίε. Πώ μπορούμε να απελευθερώσουμε το πνευματικό και να το αξιοποιήσουμε. Όμω είπαμε έχουμε αυτά τα 35 εκατομμύρια αφορούν όλη την ε, βιομηχανία. Ε, τώρα που υπάρχει κρίση, τώρα μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε. Ίσως χρειάζονται κάποια υπηρετέρα μέτρα. Με αυτά τα χρήματα μπορούμε να έχουμε κάποιο ε, μεστό περιεχομένο πρόγραμμα. Μπορούμε έτσι να έχουμε κάποια φιλόδοξα προγράμματα, αλλά έχουμε... ο περιορισμό είναι αυτό το ποσό, όπως το, το, το, πρόγραμμα για την απόσυρση των παλιών σκαφών. Πρόεδρε, απάντησα ό,τι μπορούσα, ελπίζω. Ευχαριστούμε. Ξέρω ότι ο αντιπρόεδρος Φανταλίν έχει κάτι να σας ρωτήσει, να το διευκρινίσετε. Που θα του δώσω το λόγο. Κύριε Πλάσχαρτ, ε, κύριε Κόλ, Θα λάβει μετά το λόγο. Παρακαλώ, ήταν τρίτο όμως το χρονικό όριο. Φαντάρα. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ξανατονίσω γιατί μάλλον διαφέρουμε εδώ πέρα. Έχει τελειώσει η ώρα των λόγων. Πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε γιατί πριν μιλούσαμε για τους ευρωπαϊκούς διαδρόμους, την κατάρτιση των ανθρώπων τελικά και θα φτάσουμε να εξαφανιστεί τελείως ε, η εσωτερική ναυσιπλοεία. Επίσης, τα λεφτά τα οποία υπάρχουν στον, ε, στο Ταμείο Παροπλισμού και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με τυχόν νέα μέτρα. Γιατί τι θα γίνει. Θα οδηγηθούμε σε πάρα πολύ μεγάλη χωρητικότητα του κλάδου. Πρέπει λοιπόν τι θα γίνει. Να επανεργοποιηθεί και η απόσυρση και τυχόν λεφτά από οτιδήποτε προσμό να αυξηθεί οπωσδήποτε το ποσό και βεβαίως να αποσυρθούν πρώτα απ' όλα και να φύγουν από την ε, αγορά τα πλοία εκείνα τα οποία είναι ε, παλιά και ρηπαίνουν περισσότερο. Αλλά πρώτα απ' όλα να προλάβουμε να κάνουμε κάτι όσο υπάρχει ακόμα κλάδος. Η κυρία Βόρτμαν Κόλ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ ρώτησα πότε αυτή η ομάδα εργασίας θα καταλήξει σε κάποια συμπεράσματα και πότε αυτά τα συμπεράσματα μπορούν να υποβληθούν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Διότι το μήνυμα είναι σαφές. Θέλουμε να βοηθήσουμε και να υπάρχουν μέτρα τα οποία να είναι σαφή. Όμως αυτή η ομάδα εργασίας πότε θα καταλήξει σε κάποια συμπεράσματα. Κύριε Πακέ. Ευχαριστώ. Εάν συμφωνείτε μπορούμε να συζητήσουμε την προσέγγιση σας περαιτέρω. Όμως το να συνδυάσουμε τους παλιούς και τους καινούριους κανόνες ε, υπάρχει ένα πρόβλημα. Δεν υπάρχουν... Ε, το πρόβλημα είναι με την απόσυρση που, που προτείνεται. Πού θα βρούμε τα καινούργια πλοία. Δεν υπάρχουν καινούργια πλοία. Υπάρχουν κάποια ε, πλοία τα οποία έχουν παραγγελθεί, τα οποία θα έρθουν και τα οποία όμως δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο οποιοδήποτε μέτρου. Ε, άρα θα, έχει, θα υπάρχει απόσυρση ή παροπλισμός από μόνος του. Δεν θα υπάρχει σαν ε, κομμάτι ενός ε, ευρυτέρου προγράμματος. Τώρα, τα πάντα δεν εξαρτώνται από αυτήν την ομάδα εμπειρογνωμόνων που θα συγκληθεί και που θα συζητήσει και με τον Επίτροπο κύριο Κάλλας τον Φεβρου... εμείς αποφασίσαμε ε, ε, ε, ότι με τις Ολλανδικές Αρχές θα ολοκληρώσουμε την μελέτη του προγράμματός τους τον Φεβρουάριο, όμως και η Ολλανδική Κυβέρνηση δεν έχει ολοκληρώσει το... την ανάλυση του προγράμματος. Περιμένουμε να οριμάσει και το πρόγραμμα των Ολλανδών ε, γιατί θα είναι ένα ε, πολύ σημαντικό κομμάτι, μια σημαντική συνιστόσα της γενικότερης ευρωπαϊκής ε, προσέγγισης. Λοιπόν, επειδή η κατάσταση πιέζει, τα πράγματα είναι σοβαρά, έχουμε βάλει ένα ε, χρονοδιάγραμμα, τον Φεβρουάριο. Βέβαια, τα πάντα εξαρτώνται και όλες και από το ε, πότε θα έχουμε στη διάθεσή μας και την, ε, το Ολλανδικό σενάριο, αν θέλετε. Και θα επανέλθουμε σε εσά. Καλώς λέει ο Πρόεδρος. Θα, θα το έχουμε από κοντά, αν θέλετε, το όλο θέμα. Θα το παρακολουθούμε Μέχρι τώρα δεν είχαμε δώσει την δέουσα προσοχή στο πρόβλημα των εσωτερικών, της εσωτερικής ναυσιπλοείας. Ε, τώρα νομίζω ότι θα πρέπει να ασχοληθούμε πολύ συγκεκριμένα. Λοιπόν, περνάμε στο επόμενο σημείο. Το θέμα είναι η έκθεση της κυρίας Βλάστο, ε, την λευκή Βίβλωση για τις κλιματικές αλλαγές. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε, συγγνώμη. Καταρχάς ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους που βοήθησαν ε, στην σύνταξη της έκθεσης. Ε, έχουμε 38 τροπολογίες. Θα μιλήσω μόνο για τις τροπολογίες που γίνονται δεκτές. Υποστηρίζω όλες τις προτάσεις που βελτιώνουν να κατανοήσουμε καλύτερα τα αποτελέσματα των κλιματικών αλλαγών, διότι μόνο εάν κατανοήσουμε όλα αυτά τα περίπλοκα φαινόμενα θα μπορέσουμε να προσαρμόσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την, ε, τις μεταφορές ε, και τον τουρισμό. Γι' αυτό ακριβώς θα πρέπει να, να βελτιώσουμε την ανταλλαγή καλών ε, πρακτικών και εμπειριών στον τομέα αυτό. Θεωρώ επίσης ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να ζητήσουμε από την Κομισιό να υιοθετήσει μια ολοκληρωμένη και συστημική ε, προσέγγιση του προβλήματος, διότι το πρόβλημα αυτό πρέπει, δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο από, την, από τον τομέα των μετηφορών. Θα πρέπει να, να το εξετάσουμε και από τη σκοπιά της δημόσιας υγείας, της ενέργειες της χωροταξικής πολιτικής. Δεν πρέπει να ξεχνάμε επίσης και τις ζώνες της ε, Ευρωπαϊκής Επικράτειας που είναι ευάλωτες, παραδείγματος χάρη οι περιοχές, οι παράκτιες περιοχές, ε, διότι η ευαισθησία τους θα επιδεινωθεί λόγω ακριβώς των κλιματολογικών αλλαγών και δεν πρέπει να, να αγνοούμε ότι θα υπάρξουν και οικονομικά προβλήματα τα οποία θα επιδεινωθούν. Γι' αυτό θα πρέπει να βοηθήσουμε όλους τους οικονομικούς παράγοντες αυτών των ευάλωτων ζωνών. Θα ήθελα να επιμείνω στο γεγονός ότι με τις κλιματικές αλλαγές θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τον τομέα των μεταφορών στο σύνολό του χωρίς να ξεχνάμε κανένα, κανένα μέσο μεταφοράς. Με, με κάποιους συναδέλφους μπόρεσα να καταλήξω σε κάποιους συμβιβασμούς. Το βασικό σημείο πάνω στο οποίο συμφωνήσαμε είναι το εξής. Είναι ουσιαστικό να βελτιώσουμε σημαντικά τις ε, επενδύσει όσον αφορά την τεχνολογία και την έρευνα έτσι ώστε ε, να μπορέσουμε να προσαρμόσουμε την τεχνολογία στις κλιματικές αλλαγές. Αυτός ο συμβιβασμός δημιουργεί, δημιουργεί αν θέλετε μία νέα παράγραφο και πιστεύω ότι οι δαπάνες θα πρέπει να κινητοποιηθούν έτσι ώστε να περιορίσουμε τους παράγοντες που προκαλούν εν μέρη αυτές τις κλιματικές αλλαγές. Πιστεύω δηλαδή ότι θα πρέπει να υποστηρίξουμε την ε, ανάπτυξη καθαρών αυτοκινήτων, την, ε, την ε, προώθηση μέσων μεταφοράς εφιών και αυτό ανεξάρτητα από το τι μέσο μεταφοράς, οδικό, ένα αέριο, σιδηροδρομικό, θαλάσσιο κτλ. Επίσης, ε, οι τροπολογίες 11 και 14 ε, που ε, γίνονται δεκτές για το, που αφορούν το αστικό περιβάλλον. Επίσης, πιστεύω ότι θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν μιλάμε για για την προσαρμογή των χρηματοδοτήσεων που αφορούν τις κλιματικές αλλαγές. Η Κομισιόν έπρεπε να βρει κάποιες καινοτόμες, ε, καινοτόμους τρόπους ε, χρηματοδότησης. Η άποψη που είχε εκφράσει τότε δεν είναι δεκτή από όλους τους συναδέλφους. Συζητώντας όμως μαζί τους, σκέφτηκα κι εγώ και βρήκα ένα συμβιβασμό που διευκρινίσει σαφέστατα ότι ο την αρχή του ότι ο Ριπένων πληρώνει. Θα πρέπει η Κομισιόν βέβαια να συμπληρώσει αυτή τη χρηματοδότηση χρησιμοποιώντας πόρους από τα διαρθρωτικά ταμεία και από το πρόγραμμα οικονομικής ανάκαμψης. Οι επιχειρήσεις αυτές από πλευρά τους θα πρέπει για όλους τους τύπους μεταφορών να εντάξουν το εξωτερικό κόστος το οποίο αφορά τις κλιματικές αλλαγές. Αγαπητοί συνάδελφοι, αυτό ήθελα, αυτά ήθελα να πω όσον αφορά ε, τις τροπολογίες που μας έχουν ε, υποβληθεί. Θα πρέπει βέβαια να συζητήσουμε μαζί και κάποια άλλα σημεία ε, τα οποία παραμένουν σε κρεμότητα, ή τα διαφωνούμε. Να ολοκληρώσω όμως λέγοντας ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό η Επιτροπή μας να υιοθετήσει μια σαφή στάση πάνω σε αυτό το θέμα μίζωνος σημασίας που θα έχει ε, πολύ σοβαρές συνέπειες ε, στην πολιτική μεταφορών. Ε, συνάντησα τον συνάδελφο Βιτόριο Πρόντι, ο οποίος είναι εισηγητής στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, που εκείνη είναι η καθήλυνα αρμόδια επιτροπή και μου είπε ότι συμμερίζεται κάποιες από τις ανησυχίες μας. Όμως, επέμενε ο κύριος Πρόντι, ότι θα πρέπει η η έκθεσή του να περιοριστεί μόνο στις ε, ε, κλιματικές αλλαγές και δεν θα ε, συζητήσει για τα μέτρα καταπολέμησης των κλιματικών αλλαγών. Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να καταβάλουμε μια προσπάθεια στην γνωμοδότησή μας έτσι ώστε η πρότασή μας να υιοθετηθεί. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σίμψον. Σας ευχαριστούμε αγορητές έχουν γραφεί στο κατάλογο οπότε. Να δούμε τι θα γίνει γιατί μας πιέζει ο χρόνος. Α, 8. Και ξεκινούμε με τον ε, κύριο Γκρός. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Πρώτα πρώτα ευχαριστώ την συγκεντρία για το κείμενό της και ευχαριστώ τους συναδέλφους για την συμβολή τους τη συμβολή του το να καταφέρουμε να συμβαστούμε σε ορισμένα ζητήματα. Θα πρέπει επίση να δούμε τι γίνεται όσον αφορά την ανάπτυξη, την αλλαγή του κλίματος. Πάρα πολλές φορές ε, αναφέρονται με αυτά τα προβλήματα ε, οι μεταφορές, ε, αλλά ποτέ δεν, δεν, δεν ζυγίζεται, δεν, δεν εκτιμάται στο σύνολο στο σύνολό του το, το, το, θέμα, το πόσο σημαντικό είναι και θα πρέπει όμω τώρα να δούμε μια που είμαστε η κυρίω αρμόδια επιτροπή να δούμε πώ η γνώμη μας θα ληφθεί υπόψη. Δεν είναι να λέμε ότι 25% των εκπομπών προέρχονται από τι μεταφορέ και κατόπιν να σταυρώνει κανεί τα χέρια του. Επομένω, ε, εφόσον υπάρχουν οι πόροι, θα πρέπει να, να δούμε πώ θα κάνουμε κάτι παρά την οικονομική κρίση. Γιατί είπαμε, έχει σημαντικό ο κλάδο, αλλά θα πρέπει να διπλικοδείται όπω πρέπει επίση. Θα πρέπει να βλέπουμε και πλευρά τη ενεργειακή πολιτική τι γίνεται. Είναι κάτι το οποίο εδώ πέρα έχει ζητηθεί στο παρελθόν. Να σκρεβέτσω τη θέση του ΕΛΚ. Θα πρέπει να δημιουργήσουμε κάποια κίνητρα. και να γίνεται η κατασκευή σκαφών με τέτοιο τρόπο, το ώστε να, μην, να είναι φιλική στο περιβάλλον. Επίσης, ο Μουλίνο να πληρώνει. Το σημαντικό βέβαια δεν είναι το ποιο πληρώνει. Το θέμα είναι να χρησιμοποιήσουμε ε, ε, του πόρου που έχουμε για να μειωθεί η μόλυνση. Αυτά θα συζητούμε πρόσφατα και ξέρουμε ότι γίνεται να έχουμε μια καλύτερη κατανομή του κόστους. Αυτά συνάδελφοι και σας ευχαριστώ για τη συνεργασία σας. Εμείς ευχαριστούμε κύριε συνάδελφε, κύριε συναλόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, δεν θα με γρηγορήσω. Και πρώτα πρώτα θα ήθελα να σας πω ότι ευχαριστεί η πολιτική μας ομάδα την εισηγήτρια για την έκθεσή της, τη μελέτησε και τις 38 μας τροπολογίες, γιατί κατέβαλε προσπάθειες να, να τα βρούμε. Και επίσης θα πρέπει να πούμε ότι είναι πάρα πολύ θετικό ότι περισσότερες από τις τροπολογίες εκείνες θεωρήθηκε ότι συνάδουν προς τις απόψεις της εισηγήτριας. Επομένως, η πολιτική μας ομάδα δεν μπορεί παρά να επιψηφίσει αυτήν την έκθεση. Τώρα, σαν να τις επιμέρους προτάσεις, επίσης θεωρούμε θετικό ότι γίνεται αποδεκτή η αρχή του ότι ο Μιλήνων πληρώνει και σε πολλές από αυτές τις προτάσεις διαπιστώνεται το πόσο σημαντικό είναι το να υπάρξουν επενδύσεις στις ε, υποδομές, το να υπάρχει ευελιξία και να υπάρξει καινοτομία, να υπάρξει κινητικότητα σε σχέση με τις πόλεις, η οποία να είναι βιώσιμη. Και να δούμε τι θα γίνει με τις πάρα πολύ ευαίσθητες, δύσκολες ε, περιοχές. Τις παράκτιες και τις ορεινότερες. Αυτές οι δύο κατηγορίες περιοχών θα πρέπει να προσεχθούν σε σχέση με την αλλαγή του κλίματος. Τέλος, συμφωνώ με τις τεχνικές ε, αλλαγές ε, που έχουν προταθεί. Εμείς σας ευχαριστούμε. Κύριε Πρόεδρε, τελευταία φορά που συνδίκαμε, ξανασυζητήσαμε το θέμα αυτό δηλαδή το ότι οι μεταφορές ακόμα δεν έχουν διδραματίσει πλήρως το ρόλο τους. Οπότε πάρα πολύ σωστά είναι αυτά το οποίο αναφέρθηκαν και πάρα πολύ θετικό το ότι πετύχαμε αυτό το συνδυασμό Και επίσης θεωρούμε ότι καταφέραμε να βρούμε μια πιο ευστοχή λύση, ιδίω όσον αφορά την εσωτερήκευση των, του, του κόστου των δαπανών. Μεταφορές και τουρισμός. Γιατί θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη των κλαδών μεταφορών πάντα. Και κάθε φορά να τονίζετε πόσο σημαντική είναι η εσωτερική αγορά για την Ένωση. Είναι το ίδιο σημαντική όσο και η προστασία του περιβάλλοντος. Και να δούμε τι είδους εγγυήσεις θα παρασχεθούν στο μέλλον για τις μεταφορές. Θα πρέπει βεβαίω να συγκρατήσουμε τη μόλυνση, θα πρέπει να δούμε πώς ο κλάδος δεν θα συμβάλλει τόσο πολύ την αύξηση της ε, μόλις ατμόσφαιρας. Γι' αυτό και σας λέω ότι οι επιτευθέντες ε, συνέβασμοί είναι πάρα πολύ θετικοί. Ο επόμενος. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Τους πράσινους δεν μπορέσα, εμείς οι πράσινοι μάλλον, δεν ε, πήραμε μέρος στην ε, διαμόρφωση του συμβιβασμού. Και ίσως είναι δικό μας το πρόβλημα, δεν ξέρω, αλλά τέλος πάντων, ε, τι να πω, δεν λειτουργήσε καλά η συνεργασία στο εσωτερικό του Κοινοβουλίου. Διάβασα όμως το κείμενο και δεν μπορώ να καταλάβω τι θα γίνει, πώς θα ψηφίσουμε. Υπάρχουν προφορικές τροπολογίες που είναι πολύ γενικές, θα έλεγα. Στο σύνολο της αυτή η έκθεση αφορά μια κάποια προσαρμογή. Μου έκανε εντύπωση όταν άκουσα ότι ο κύριος Πρόντι είπε ότι δεν θα έπρεπε να ασχοληθούμε εδώ με λύσεις, δηλαδή με την μείωση της μόλυνσης ε, ε, που προκαλεί το διοξίδιο του άνθρακα που προκαλούν οι μεταφορές. Θα ασχοληθούμε ή δεν θα ασχοληθούμε τελικά. Γιατί θα πρέπει να ασχοληθεί και η Κομισιόν και με τη συνεισφορά, αν θέλετε, της, του τομέα των μεταφορών. Ε, τη συνεισφορά στις κλιματικές αλλαγές. Δεν μπορούμε να περιμένουμε Δεν μπορούμε να περιμένουμε ε, να έχουν πλημμυρίσει, να, να έχουν λιώσει οι πάγοι, να, έχει πλημμυρίσει, να έχουν πλημμυρίσει οι δρόμοι και τα αυτοκίνητα αντί για να χρειάζονται ε, φλωτέρ για να μετακινηθούν. Τέλος πάντων, οι τροπολογίες που έχουμε υποβάλει έχουν σαν στόχο να βελτιώσουν τη συνεισφορά μας, έτσι ώστε να μειωθεί η μπόλυνση του περιβάλλοντος. Ελπίζω δηλαδή ότι όλες οι τροπολογίες οι οποίες αφορούν τον περιορισμό της μόλυνσης ατμοσφαιρικής ρήπανσης θα υπερψηφιστούν. Κύριε Φώστερ, ευχαριστώ Πρόεδρε. Δεν ξέρω τι θα γίνει στην Επιτροπή Περιβάλλοντος βέβαια και τι θα βγει, αλλά νομίζω ότι η κυρία Βλαστό προσπαθεί να αντιμετωπίσει ρεαλιστικά το πρόβλημα. Είμαστε η Επιτροπή Μεταφορών. Τι μεταφορέ τι χρειαζόμαστε, παρόλο το ότι έχουν διάφορα κακά. Αλλά τέλο πάντων πιστεύω ότι θα πρέπει να βρούμε ε, κάποιες συμβαστικές ε, προτάσεις. Ή τις τροπολογίες θα πρέπει να τι μελετήσουμε. Αλλά πιστεύουμε ότι τις περισσότερες από τις ε, τροπολογίες που, ε, πρότεινε η κυρία Βλαστό μπορούμε να τις δεχτούμε, εκτός από τρεις-τέσσερις θα πρέπει να τονίσουμε και την, ε, τον ιδιαίτερο χαρακτήρα των ορεινών περιοχών και όλα αυτά. Αλλά τέλος πάντων, ε, σε αυτό το στάδιο ε, πιστεύω ότι θα, την, θα υποστηρίξουμε την γνωμοδότηση, την έκθεση. Τώρα βέβαια θα πρέπει να δούμε τι θα, πώς εξελιχθούν οι συζητήσεις. Αυτό το οποίο μας ανησυχεί όμως λιγάκι είναι η αλλαγή της διατύπωσης σε κάποιο σημείο. Μιλάμε για από global warming, από ε, παγκόσμια θέρμανση, η θέρμανση του πλανήτη, μιλάμε, σε μιλάμε για κλιματικές αλλαγές. Και ένα στοιχείο το οποίο έθιξε η συνάδελφος είναι η ρήπανση, η μόλυνση. Και πιστεύω ότι ο όρος αυτός pollution είναι πάρα πολύ σημαντικός στην συζήτηση. Και πρέπει να γίνουν και κάποιες έρευνες ε, και στον τομέα των μεταφορών έχουμε επενδύσει τεράστια ποσά στις, ε, στην έρευνα. Το πρόβλημα είναι ότι τα επόμενα δύο χρόνια όλοι θέλουν έρευνα σε όλους τους τομείς. Άρα πρέπει να είμαστε κάπως ρεαλιστές. Γι' αυτό θα πρέπει να το ζητήσουμε το θέμα και η ομάδα μας ούτως ή άλλως υποστηρίζει τις περισσότερες τροπολογίες της κυρίας Βλαστό. Τώρα βέβαια δεν υποστηρίζουμε για κάποιες άλλες, αλλά τέλος πάντων. Τι, όταν ψηφίσουμε την Πέμπτη θα έχουμε πάρει και την απόφασή μας. Τετάρτη ψηφίζουμε, Τετάρτη απλώς να σου το υπενθυμίσω. Η κυρία Γιάλα Σέντερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. όλα σας ευχαριστώ σας και ιδιαίτερα στην ε, κυρία Βλαστό για την γνωμοδότηση. Και ήταν πάρα πολύ σωστή η συνεργασία και με τους επιμέρους προτείναντες της τροπολογίας αλλά και με τον εισηγητή στην Επιτροπή Περιβάλλοντος. Πάρα πολύ σωστή η διαδικασία αυτή γιατί όταν έρθει η ψηφοφορία ε, δεν χρειάζεται τίποτα επαναστατικέ διαδικασίε. Χρειάζεται να έχει υπάρξει προηγούμενη διαπραγμάτευση με τον εισηγητή και με την ε, ε, αρμόδια ή συναρμόδια επιτροπή. Οπότε πάρα πολύ καλά τα πήγε και προ τα δύο μέτωπα εισηγητή. Όσον αφορά τώρα τον συμβασμό αυτών, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Ε, τον ευχαριστώ για, για, το, για το ότι δεν σήμερα με τι τροπολογίε μου. Όμω το μόνο που θα ήθελα να πω και να ζητήσω από, τον εισηγητή, από την εισηγητή κάτι το οποίο αφορά τη, τη, το, το γάμα, τη, τη συμβαστική γάμα. Εκεί που είναι ουσιαστικά και πρόταση και τροπολογία αυτό που προτείνει ο κ. Χαντράουι. Οπότε, ερωτώ, με, με αυτήν την τροπολογία θα συμφωνούσατε ε, να διατυπώσουμε ακριβώς ενώ αυτή της αρχής ότι όποιος ε, μολύνει πληρώνει, ο Ριπένον πληρώνει, να δούμε πώς θα γίνει αυτό πιο εύχριστο ο ε, ως ρύθμιση για όλους, όλα τα είδη μεταφοράς. Στα πλαίσια της προσπάθειας που κάνουμε να είναι πιο εύρυθμη η λειτουργία του κλάδου, ε, του κλάδου των, των, των μεταφορών. Και έτσι συνενετικά να περάσει αυτή η τροπολογία, χωρίς να αντιπαρατεθούμε. Να δούμε και ποιος είναι ο κοινωνικός αντίκτυπος μιας τέτοιας ρύθμισης. Μια που γενικότερα στα πλαίσια της πράσινης απασχόλησης υπάρχουν τέτοιου είδους ε, θετικοί κοινωνικοί αντίκτυποι, κοινωνικά, κοινωνικές συνέπειες πρόληψη είναι το κλειδί για την αντιμετώπιση της παραδείγματος του περιβάλλοντος βέβαια και γι' αυτό και είναι θετικό το ότι έχει πρωτοπόρο σχέση με αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση όμως θα πρέπει κανείς να προσαρμόζεται οπότε χρειάζεται και αυτό αφορά και την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και τα κράτη-μέλη σε σχέση όμως και με τις τρίτες χώρες. Ποτέ δεν εργάζεται να προσαρμοστεί κανένας επομένως. Θα πρέπει κάποια στιγμή να το ζητήσουμε ακριβώς αυτό το, το ζήτημα το συγκεκριμένο το, της προσαρμογής. Ε, ευχαριστώ και ο Πρόεδρος. Μια... Η περιγραφή του προβλήματος δεν το λύνει και ένα σχέδιο δεν είναι δράση. Και αυτό λείπει εδώ πέρα από αυτή την έκθεση. Στην αρχή αναφέρεται πως η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμευτεί να μειώσει κατά 20% τις εκπομπές μέχρι το 2020. Ωραίο σχέδιο. Ίσως το πετύχουμε, ίσως όχι, αλλά ένα είναι σαφές, χωρίς ριζική αλλαγή των συγκοινωνιών δεν θα το καταφέρουμε. Εκεί πέρα παράγεται σχεδόν 30% ε, των εκπομπών και από το 1990 έχουμε αύξηση 35%. Σε άλλους ε, τομείς, στη βιομηχανία, π.χ. έχουν ε, υπάρξει πάρα πολύ μεγάλες επενδύσεις, όπως επίσης και στη θέρμανση των σπιτιών. Εάν θέλουμε να καταπολεμήσουμε λοιπόν την κλιματική αλλαγή και στο μέλλον, το κάναμε αυτό αλλού, τα γνωρίσαμε τελείως στην ε, συγκοινωνίε και αυξήθηκε. Αυξήθηκαν οι κομπέ. Μέχρι σήμερα δεν υπάρχει στόχος για τι συγκοινωνίε. Θέλουμε 20%, 30%, 10%, θέλουμε μια σταθεροποίηση, τίποτα. Ποτέ δεν υπάρχει στόχος. Και όποιος δεν έχει στόχο δεν μπορεί να παραπονιέται κιόλα βέβαια ότι δεν επέτυχε τον στόχο. Απλό αυτό, αλλά δεν βοηθάει την κλιματική αλλαγή. Γι' αυτό θέλω να ξαναρωτήσω γιατί κάνουμε το λάθος της Κομισιόν που δεν είναι καν σε θέση να ορίσει ένα στόχο. Αρνήθηκε να απαντήσει ο υποψηφίο επίτροπος όταν τον ρωτήσαμε εάν πρέπει να έχουμε δεσμευτικό στόχο για τι συγκοινωνίε. Το Γερμανικό Ομοσπονδιακό Συμβούλιο το αποφάσισε ομόφωνα. Δεν μιλάμε και για κανένα πράσινο. Δεν υπάρχει πράσινο μέλος εκεί πέρα. Να υπάρξει συγκεκριμένα δεσμευτικό στόχος 20% μέχρι το 2020. Ναι, συναπόφαση ήταν και δική σας. Και τώρα καθόμαστε εδώ πέρα και δεν λέμε στόχο. Χρειαζόμαστε ένα στόχο για να καταπολεμήσουμε την κλιματική αλλαγή. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Τίκαν. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Θα ήθελα να συγχαρώ την κυρία Βλαστό για την ε, γνωμοδότησή τας. Εδώ είπαμε ότι θα πρέπει να προσαρμοστούμε στις κλιματικές αλλαγές. Όταν μιλάμε για προσαρμογή θα πρέπει να μιλάμε επίσης και για την πρόληψη από, πλημέ, και το πρόγραμμα Γαλιλαίο και ε, είναι, παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Επίσης και όλα τα μέτρα τα οποία πρέπει να ληφθούν για την διαφύλαξη των σοβαρών έργων υποδομής. Εμείς έχουμε ζητήσει οι θαλάσσιες μεταφορές να αποτελούν ένα κομμάτι του συστήματος ETS. δηλαδή του συστήματος εμπορίας ε, εκπομπών. θα πρέπει να ε, ολοκληρώσουμε την, το, όλο, το όλο πρόγραμμα συζητώντας επίσης και καθορίζοντας και την, τους διαδρόμους για τις μεταφορές ε, των εμπορευμάτων όπως επίσης και την, τις ε, ταχύες σιδηροδρομικές μεταφορές. Το πρόβλημα ποιο είναι όμως ότι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε ευφυή, e e, έξυπνα δηλαδή μεταφορικά μέσα, έτσι ώστε να περιορίσουμε τις ε, εκπομπές ε, των αερίων και να περιορίσουμε την μόλυνση και τη ρήπανση. Ευχαριστώ ε, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Βλαστό για τη γνωμοδότησή της, ε, διότι στην ε, έκθεση αυτή υπάρχουν πάρα πολλά ενδιαφέροντα σημεία τα οποία συμμεριζόμαστε όλοι. Όμως για την αρχή ας πούμε ο Ριπένων πληρώνει. Είναι μια αρχή που εμείς υποστηρίζαμε εδώ και πολλά χρόνια, ετία, και χαίρομαι που συμπεριλαμβάνεται στην έκθεση αυτή. Τώρα, παρά τις ε, τεχνολογικές ε, προόδους ε, δεν έχουμε, δεν έχουμε μπορέσει να περιορίσουμε τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Ε, και υπάρχουν ε, τα θέματα αυτά θίγονται και στις διάφορες τροπολογίες που έχουν υποβληθεί. Η έκθεσή μας όμως, η έκθεση αυτή συγκεκριμένα αναφέρεται στην αδυναμία μας να προσαρμοστούμε στην κοινωνία του 21ου αιώνα. Κοινωνία δηλαδή τη σημερινή, αύριο, ε, του αύριο. Και δεν θα πρέπει να μιλάμε μόνο για τις παράκτιες ή τις ορεινές περιοχές, αλλά και για τις πόλεις μας. Οι πόλεις μας που υποφέρουν από κυκλοφοριακή συμφόρηση και πόλεις που κάνουν τη ζωή των πολιτών ανυπόφορη. Επομένως θα πρέπει να ε, προχωρήσουμε ας πούμε σε κάποιες ριζοσπαστικές αρχές π.χ. να έχουμε ένα αυτοκίνητο το οποίο αποτελεί αντικείμενο ε, μοιρασιάς δεν, να μην έχουμε αποκλειστικά δικαιώματα ε, δηλαδή δικαιώματα αποκλειστικής ιδιοκτησίας πάνω σε ένα αυτοκίνητο θα πρέπει να δούμε το μέλλον και να, έχουμε, να καταλήξουμε σε ένα πακέτο αν θέλετε συνολικό για τις, ε, μεταφοράς, ε, για τις μεταφορές και να μην τα βλέπουμε μεμονωμένα κάθε μέσο μεταφοράς αλλά να το δούμε σφαιρικά και να συζητήσουμε και τα θέματα και των, των επενδύσεων και των χρηματοδοτήσεων κτλ. Ο κύριος Ντελσάλεξ, Ο ονόματος της Κομισιού, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Βλαστό αλλά και τα άλλα μέλη της Επιτροπής Μεταφορών για τις τροπολογίες ε, που υπέβαλαν Ελπίζω ότι η γνωμοδότηση θα γίνει, θα ληφθεί υπόψη στην ε, έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος έτσι ώστε να ε, τονιστεί και η σημασία που έχει ο τομέας των μεταφορών στο όλο θέμα των κλιματικών αλογών διότι αυτός ο τομέας μέχρι τώρα δεν είχε αποτελέσει αντικείμενο μιας ιδιαίτερης προσοχής σε σχέση με άλλους τομείς όπως είναι η γεωργία ή η υγεία. Ε, εκεί είχαν γίνει αναλύσεις ε, πιο προχωρημένες. Λοιπόν, συμμεριζόμαστε και συμφωνούμε με την, ε, με την άποψη που ακούστηκε ότι η έκθεση δηλαδή θα πρέπει να εστιάσει περισσότερο στα σημεία προσαρμογής διότι υπάρχουν και κάποια κομμάτια του κειμένου της Κομισιόν που έχουν λάβει υπόψη ε, τα θέματα μετριασμού των κλιματικών ε, αλλαγών που θα μπορούσαν να προέλθουν από τις μεταφορές. Ε, πιστεύουμε ότι οι συμβαστικές τροπολογίες θα μπορούσαν να αποτελέσουν μια γέφυρα με, αυτή την, με αυτό το μετριασμό των κλιματικών αλλαγών και να τονίσουμε ότι μπορούμε να λάβουμε υπόψη μας ε, την επίτευξη των βιώσιμων στόχων στον τομέα των ε, μεταφορών, ε, υιοθετώντα και την αρχή του ορυπαίνων πληρώνει. και μπορούμε να προχωρήσουμε σε έναν, σε εξυγχρονισμό των, των επενδύσεων. Θα πρέπει να ε, δούμε πώς θα προσαρμοστούν οι διάφορες πολιτικές και η πολιτική μεταφορών και αυτές οι προσαρμογές θα ε, συμπεριληφθούν σε, μια, ένα επόμενο κείμενο της Κομισιόν, στην Λευκή Βίβλο για, τα, για, τις, για την πολιτική μεταφορών, για το 8ο πρόγραμμα πλαίσιο και προσπαθούμε να προωθήσουμε και την ε, καλύτερη χρήση των υπαρχών των μέτρων, π.χ. πούμε των διορθωτικών ταμείων, έτσι ώστε βραχυπρόθεσμα να μπορέσουμε να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα και θα συνεργαστούμε με τη Γραμματεία της Επιτροπής Επιτροπή Μεταφορών έτσι ώστε να ολοκληρωθεί η γνωμοδότηση και η γνωμοδότηση αυτή να αντικατοπτριστεί και στη γνωμοδότηση τη Επιτροπής Περιβάλλοντος. Ευχαριστώ κύριε Ντελσάλα ή η η κυρία Βλαστό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δύο δευτερόλεπτα μόνο. Θα ήθελα να επαναλάβω στους συναδέλφους ότι ε, μπορεί να μην συμφωνούμε, όμως εδώ δεν μας ζητήθηκε στην έκθεση αυτή να μιλήσουμε για την καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών. Ε, και ο κύριος Πρόντι μας, ε, μου το είπε, μου το διευκρίνησε ότι μπορεί να μην, να μην συμφωνούμε, όμως αυτό το οποίο αναφέρει η Λευκή Βίβλος είναι η προσαρμογή στις κλιματικές αλλαγές και κανείς δεν μου ζήτησε να έρθω σε επαφή μαζί σας για να συζητήσουμε τις ε, προσαρμογές των τροπολογιών που υποβάλλατε εσείς. Λοιπόν, για την τροπολογία 4 γι' αυτό είπα ότι θα πρέπει να μιλήσουμε για όλες τις μεταφορές και να μην μιλήσουμε μόνο για το σιδηρόδρομο και τα αυτοκίνητα. Αυτά ήθελα να πω για τον τουρισμό. Προφανώς ε, ο τουρισμός έχει κάποια σημασία, έχει τη σημασία του και ο τουρισμός συνδυάζεται με τις μεταφορές ούτως ή άλλως, άρα δεν μπορούμε να τον διαφοροποιήσουμε. Αυτά είχα να πω κύριε Πρόεδρο. Ευχαριστώ κύριε Βλαστό. Να σας υπενθυμίσω, επειδή αλλάξαν ημερομηνίε, θα ψηφίσουμε την Τετάρτη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπορούμε να περάσουμε τώρα στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης, που είναι δική μου έκθεση. για, την, ε, για μια τεχνική ε, ε, τεχνικό κείμενο κύριε, που αφορά τους κοινωτικούς προσανατολισμού για την ανάπτυξη του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών. Πρόκειται για μια αναδιατύπωση. Είχα μια άτυπη συνεδρία, ανεπίσημη συνάντηση με τους σκιώδεις εισηγητές για να δούμε αν μπορούσαμε να καταλήξουμε σε κάποια συμφωνία. Ίσως η Κομισιόν τώρα να ήθελε, η εκπρόσωπος του Συμβουλίου θα ήθελε να πάρει το λόγο. Οι νομικές υπηρεσίες του Κοινοβουλίου με ενημέρωσαν ότι οι εργασίες διαβούλευσης ε, ε, των νομικών υπηρεσιών των τριών οργάνων ε, συμφώνησαν Η νομική υπηρεσία είπαν ότι το προτινόμενο κείμενο δεν αναφέρει καμία καινούρια αλλαγή πέραν αυτών που αναφέρονται στην πρόταση. Δηλαδή γίνεται μια αναδιατύπωση των προηγουμένων, ε, του προηγουμένου κειμένου, άρα το, ε, τα πράγματα είναι απλά. Μιλάμε για αναδιατύπωση υπάρχοντος κειμένου χωρίς ε, ουσιαστική αλλαγή. Το αναφέρω αυτό διότι υπήρχα υπήρξαν κάποιες νομικές απορίες για το κατά πόσον η διαδικασία που υιοθετήθηκε είναι σωστή ή όχι. Επομένως η νομική συμβουλή που μας δόθηκε είναι ότι τα πράγματα πάνε καλά. Το Συμβούλιο αποφάσισε, συμφώνησε επομένως με το κείμενο και ε, στις 18 Δεκεμβρίου υιοθετήθηκε το κείμενο από το Συμβούλιο Υπουργών και το Συμβούλιο δεν έκανε καμιά ουσιαστική αλλαγή στο κείμενο, κάποιες ε, αλλαγές ίσονος σημασίας στην αιτιολογική σκέψη. Και αυτό αναφέρεται στις ε, τροπολογίες και έγιναν επίσης και κάποιες ε, τεχνικές διορθώσεις στους χάρτες. αλλάξαν κάποια νούμερα, οι πόλεις, τα ονόματα των πόλεων διορθώθηκαν, τέτοιου είδους αλλαγές έγιναν η πρόταση από τεχνικής πλευράς ε, ε, αποτελεί μια αναδιατύπωση ενός νομικού κειμένου, όμως η Κομισιόν μέσω της αυτής της διαδικασίας αναδιατύπωσης κάνει κάποιες ε, αλλαγές ίσονος σημασίας. Όπως σας είπα, προσθέθηκαν οι χάρτες και των 10 καινούριων κρατών μελών μετά τις ε, διευρύνσεις και προσχωρήσεις ε, γίνεται, ε, υπάρχει και ένα παράρτημα ένα που αφορά την αλλαγή των, των χαρτών για το Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών από τα 10 κράτη από, μετά την, διευκρι... μετά την ε, διεύρυνση του 2003 έχουμε 2020 ε, αντί για 2010. Λοιπόν, έχουμε μια προσθήκη στο παράρτημα 1 για, που αφορά τον, τους χάρτες ε, για τα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επομένως, εφόσον και πολιτικά και νομικά μας, διαβεβαίωσαν ότι δεν υπάρχει πρόβλημα μπορώ να σας πω ότι συμφωνούμε με το κείμενο ε, και αυτόν τον ίσονο σημασίας αλλαγών που προτείνει το, Συμβούλιο και ε, θα ολοκληρώσουμε ε, το θέμα αυτό στην πρώτη μας ε, συνεδρίαση. Λοιπόν, εάν συμφωνήσουμε να προχωρήσουμε ως εξή, προτείνω στις 3 Φεβρουαρίου να είναι η προθεσμία για την ε, υποβολή των τροπολογιών, να το εξετάσουμε το κείμενο μέχρι τις 21 ε, του μηνός και η συζήτηση στην Επιτροπή 23 και ε, ψηφοφορία στην Ολομέλεια του Μαρτίου του Απριλίου. Τούτων λεχθέντων ε, δίνω το λόγο στα μέλη και στον κύριο Γκρός. Ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν θέλω να επαναλάβω αυτά τα οποία είπαμε ήδη. Και εμείς θεωρούμε αυτή την έκθεση τεχνική, δηλαδή ουσιαστική συζήτηση για τα διευρωπαϊκά δίκτυα θα γίνει εν καιρό και τότε θα λάβουμε και τον λόγο. Κανένα ένα πρόβλημα τις προσαρμογές και η προθεσμία 2010 που γίνεται 2020, οπότε υποθέτω πως το ΕΛΚ ε, θα υποστηρίξει πλήρως αυτή την έκθεση. Ευχαριστώ και σας ευχαριστώ που επαναλαμβάνετε ότι αυτό δεν αφορά τα δύο ευρωπαϊκά δικτύα, αφορά τις τεχνικές λεπτομέρειες. Ο κύριος Αλχαντραουή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, συμφωνώ πλήρως με τον συνάδελφο τον κύριο Γκρός, είναι τεχνικός ο φάκελος Και βεβαίω αν ήταν αλλιώ τα πράγματα θα έπρεπε να έχουμε προβλέψει και περισσότερο χρόνο από το μισάωράκι στην ημερήσια διάταξη. Όπω λοιπόν και το ΕΛΚ και εμείς ε, την στηρίζουμε και ελπίζουμε αργότερα εντό του έτου, να γίνει μια πιο αναλυτική συζήτηση για τα διευρωπαϊκά δίκτυα και το μέλλον. Ευχαριστώ κύριε Ελχαντραουή. σα διαβεβαιώνω πως εάν αφορούσε την ουσία των διευρωπαϊκών δικτύων πράγματι θα ήταν πάνω από μισή ώρα στο πρόγραμμα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Συμφωνώ απόλυτα με αυτά που είπατε όσον αφορά την έκθεση. Επομένως, ας αναβάλουμε, την, ε, τη συζήτηση επί της ουσίας. Μιλάμε για το τέλος του 2010 για την παρουσίαση της από πλευράς της ε, Κομισιόν Ίσως θα μπορούσαμε να απευθύνουμε μία πρόσκληση προς την Κομισιό να επιταχύνει κάπως τις διαδικασίες και να ε, μας υποβάλει ένα κείμενο όσο να τον πιο γρήγορα για να το συζητήσουμε. Ο κύριος Κράμερ. Ναι, επειδή είναι τεχνική έκθεση, νομίζω υπάρχει εύκολα συνένεση. Αν ήταν επί της ουσίας, θα διαφέραμε, αλλά εδώ πέρα βεβαίως συμφωνούμε. Ο πρόεδρος. Ζήλε. Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Αλλά ευχαριστώ και για αυτό το έγγραφο. Ελπίζουμε ότι και το Συμβούλιο θα συμφωνήσει, οπότε θα μπορέσει αυτή η γνωμοδότηση να διεκπαιρεθεί γρήγορα και ότι όλα θα πάνε καλά. Εμείς ευχαριστούμε. Πήρε το λόγο ο συντονιστή μου ούτω ή άλλω. Επομένω δεν χρειάζεται να προσθέσω εγώ τίποτα. Απλώ και μόνο να πω ότι αυτό αποτελεί το βασικό κείμενο πάνω στο οποίο θα στηριχθεί η συζήτηση. Ελπίζω να το πιο γρήγορα. Για να δημιουργήσουμε μια νέα πλατφόρμα που θα πρέπει να εξεταστεί ιδιαίτερα προσεκτικά με βάση αυτά που έχουμε μπροστά μας. Δηλαδή θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, διότι όλα όσα είπαμε και πριν για το περιβάλλον, για το κλίμα κτλ. κτλ τα πάρα πολλά από αυτά εξαρτώνται και από την δουλειά που θα κάνουμε και για το μέλλον. Και από το ποιόν της δουλειάς που θα κάνουμε για το μέλλον δηλαδή. Επομένως θα ήθελα να έχουμε το κείμενο στον πιο γρήγορα, έτσι ώστε όσο να πιο γρήγορα να ασχοληθούμε τα θέματα αυτά, μια και σκέψη. Η κυρία Γιάλα Σέντερ. Ευχαριστούμε και που μας υπενθυμίζετε ότι το κείμενο για να ζητηθεί θα το έχουμε όταν εκπονίζει τις προτάσεις της οριστικά και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ότι αυτό απλώς είναι μια μικρή προσαρμογή. Παρακαλώ, όταν έχουμε την, την ενημέρωση. Μην ξεχνάτε τι γίνεται με τα πυρηνία, γιατί ξέρετε την τελευταία φορά, με την τελευταία, με την τελευταία προσαρμογή έγινε μια μικρή επανάσταση, εστασίασαν στη δημοκρατική, στην ε, εκλογική μου περιφέρεια. Οπότε παρακαλώ, μην ξεχνάτε όταν έρθει η ώρα του να δημοσιεύσετε το σχετικό χάρτη στο ίντερνετ. Εμείς ευχαριστούμε το πρόεδρος. Με, το οι χάρτες πάντα είναι ε, πάρα πολύ επικίνδυνοι για να εξάψουν τα πάθη. Κύριε Τικά, ευχαριστώ πρόεδρε. Όντως, μια τέτοια αναθεώρηση των ε, προγραμμάτων του 2010 που θα τύχουν προτεραιότητα είναι κάτι που το περιμένουμε πως και πως στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να δούμε τι γίνεται, τι θα γίνει με αυτούς τους χάρτες. Εγώ δε. Έχω την εξή ερώτηση. Βλέπουμε τι γίνεται στη Βαλτική όσον αφορά τα λιμάνια, στο παράδειγμα 51, βλέπουμε τι γίνεται στη Βόρειο θάλασσα, τι γίνεται με τον Ατλαντικό, βλέπουμε τι γίνεται με ε, την ε, Μεσόγειο, βλέπουμε τι γίνεται στη Δυτική Μεσόγειο, στην Ανατολική Μεσόγειο, αλλά, αλλά η Μαύρη Θάλασσα πουθενά δεν αναφέρεται παρά το ότι η Βουλγαρία και η Ρουμανία ε, αναφέρονται βέβαια. Αναφέρονται επομένω οι λιμένε, αλλά όχι στο χάρτη. Επομένω, νομίζω ότι θα πρέπει να προβούμε σε κάποια διόρθωση. Διότι από πλευρά Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτοί οι διάδρομοι έχουν λησμονηθεί. Δεν αναφέρονται δηλαδή μαζί με τους υπόλοιπους λιμένες της ε, Ένωσης Πασκουά. Είναι τεχνική αυτή η έκθεση και όπως όλοι συμφωνούμε πίσω από, την τεχνική, από το τεχνικό κείμενο κρύβεται ένα πολιτικό κείμενο με πάρα πολύ σημαντικές αποφάσεις. Άρα το κατώ που έχουμε να κάνουμε εδώ πέρα είναι το νωρίτερο δυνατόν σε πρώτη ανάγνωση να δούμε αυτό το κείμενο και ούτως ώστε να μην δώσουμε δηλαδή ούτε για Τεχνικέ προφάσεις, ούτε για πολιτικές ε, ε, προφάσεις, τόσο ώστε να μην τηρηθούν κάποιες δεσμεύσεις που έχουν γίνει. Άρα, να προωθηθεί, να διεκπληρωθεί το κείμενο όσο γίνεται γρηγορότερα. Σίμψον, έτσι, έτσι είναι. Α, κύριε Πακέ, τώρα σε εσά πάλι σκητάλα για ένα θέμα που είναι λιγότερο καυτό από ότι η ιστορική ναυσιπλοεία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ ε, και τον εισηγητή, ευχαριστώ και του συνάδελφου που έλαβαν τον λόγο. Γιατί Όντω, ε, καλά τα είπαν όσον αφορά το ότι θα πρέπει και να κάνουμε σε πρώτη ανάγνωση. Ναι, εδώ έχουμε μια κωδικοποίηση. Και με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να έχουμε ε, να προλιάνουμε τον δρόμο τόσο ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε προς την χάραξη πολιτική το 2010 και κατά αυτόν τον τρόπο να μπορέσουμε ε, με την συνήθεια τακτική νομοθετική διαδικασία να προχωρήσουμε με το Κοινοβούλιο να συνομοθετεί ο συνήθως. Και μην αναφέρεται στο χάρτη στα σχετικά παραδείγματα. Η Μαύρη Θάλασσα δεν υπάρχει πρόβλημα, τα προγράμματα περιέχονται, καλύπτονται, θα τρέξουν στα πλαίσια τη νέα πολιτική. Θα σα καλύψει το νέο, θα σας καλύψει το νέο πλαίσιο, μην ενισχύετε. Σίμψον. 3 Φεβρουαρίου είναι η λήξη της προθεσμίας για τις τροπολογίες σας υπενθυμίζω Πάμε τώρα στο επόμενο. Uh, το, αυτό το αυτοκόλλητο, η ευρωπαϊκή βινιέτα. Θα θυμάστε τι αποφάσισαν οι συντονιστές. Όσον σχετική παρουσίαση, όσον αφορά τη μελέτη, για να μπορέσουμε να ενημερωθούμε όσον αφορά τις τελευταίες εξελίξεις. η 10η Γενική Διεύθυνση προέβη εις αυτήν την μελέτη όσον αφορά την αναθεώρηση της ε, οδηγίας 62 του 99. Ε, τη μελέτη αυτή τη ζήτησε το Συμβούλιο, τόσο ώστε να εξασφαλιστεί το ότι Ό,τι γίνει θα είναι σύντομα με την πολιτική μας. Πήγε στον ομάδα εργασία το Δεκέμβριο. Δεν είναι μόνο η ευκαιρία που είχε η Σουηδική Προεδρία κάτι να κάνει για αυτή την πρόταση. Η μελέτη έχει διανεμηθεί. Κύριος Πασκορέλη είναι εδώ για να την παρουσιάσει. Ήρθε. Όχι. Καλά, να περιμένουμε μετά λεπτά. Θα μπορούσε να γίνει, ξέρω ότι θα πρέπει να φτάσει 5 η ώρα, αλλά θα μπορούσε να το πιο νωρί, γιατί σιγά σιγά αρχίζουν να φεύγουν οι, φεύγουν οι, τα κάτι μελη Μα, ακούτε τώρα? Τώρα? Ανοιχτό ήταν. Ε, λοιπόν, να, να περιμένουμε ένα πέντε λεπτό για να έρθει ο Πασπαρίλη, εκτό εάν ε, κάποιο από την Κομισιόν συναδελφό του έχει το, το τηλέφωνο, όταν τον πάρει τηλέφωνο, να δούμε τι γίνεται. give an eight minute recess and we start again at five. Άρα σταματάμε για λίγο και ξαναρχίζουμε στις 5 ε, ώρα.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 εδώ η κουβέντα αφορά μόνο την κουβέντα τη Επιτροπή Μεταφορών και όχι τίποτα άλλο. Οπότε κύριε Πασκορέλη, μπορείτε τώρα να λάβετε το λόγο όσον αφορά την, την μελέτη για την ε, Ευρωβινιέτα. και όποιο δεν σιωπάσει θα, το σιωπήσει να τον πετάξω έξω. Γεια σα, λέει ο κύριο Πασκορέλη. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Και συγγνώμη που άρχισα, άργησα λίγο. μεγάλη μου χαρά έρχομαι εδώ στην ε, συνάντησή σας. Σας ευχαριστώ εσάς και την Επιτροπή Τραν γιατί έτσι μου δώσατε την ε, ευκαιρία να προβώ σε αυτή την παρουσίαση και να τα συζητήσουμε κάτι το οποίο αποτελεί πάρα πολύ σημαντική ευκαιρία για μας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μπορούμε να σας εξηγήσουμε την οικονομική πτυχή που κρύβεται πίσω από αυτή μας την πρόταση για να αναθεωρήσουμε την σχετική οδηγία να την στο νέο κοινοβούλιο, στη νέα Επιτροπή των Μεταφορών. Ε, Επιτροπή όπω δημορφώθηκε με τι τελευταίε ευρωεκλογέ. Έχω εδώ ορισμένε διαφάνειε, δεν τι βλέπουν οι Έλληνε διερμηνεί. Ούτω ώστε να σα πω πώ έχει το, το, το πλαίσιο, ε, το background, πριν να αρχίσουμε να συζητάμε μετά τι ε, ε, μελέτε. Παρακαλώ στην επόμενη διαφάνεια. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας τονίσω ότι η όλη αυτή η ιδέα για το αυτοκόλλητο σήμα έχει να κάνει και με την τιμολογική πολιτική για τις μεταφορές και βεβαίως και γινόμεθα στα πλαίσια της αρχής του ότι ο ρηπαίνων πληρώνει, κάτι το οποίο από την ενιαία ευρωπαϊκή πράξη ίσχυσε και ενσωματώθηκε στις ευρωπαϊκές πολιτικές από τα μέσα της πολιτικής ε, από τα μέσα της δεκαετίας του 80. Οπότε καθ' τον τρόπο προσπαθούμε να δούμε τι θα γίνει όσον αφορά το, το, κόστος των μεταφορών, το κόστος ε, το εξωτερικό και το κόστος από την μεριά των ε, υποδομών και θα πρέπει βεβαίω εδώ πέρα να ληφθούν κάποιε συγκεκριμένε ε, πολιτικέ αποφάσει σε σχέση με το τι θα καλυφθεί όσον αφορά το εξωτερικό κόστος. Είπαμε ότι ο Ρίπανο πληρώνει και θα πρέπει όσο μόνος αυτοί οι οποίοι δημιουργούν αυτήν την, ε, αυτήν την, την, την μόλυνση, αλλά αυτοί θα πρέπει να πληρώσουν και όχι ο, ο φορολογούμενος, όχι ο καταναλωτής. Αυτό το οποίο ενδιαφέρει εδώ είναι πώς θα γίνει η κατανομή ε, μέσω αυτών οι οποίοι ε, εμπλέκονται. Βλέπουμε εδώ στην επόμενη διαφάνεια ποιοι είναι οι στόχοι και ποιος είναι ο στόχος του αυτοκόλλητου αυτού σήματος σύμφωνα με την καινούργια μας πρόταση όσον αφορά το να σταματήσουν οι μεταφορές να παράγουν διοξιδιο του άνθρακος το έχετε ακούσει πάρα πολλά σχέση με τον στόχο του 2020 και σε σχέση την Λευκή Βίβλο η οποία ε, πρόθεσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό είναι το πίνδρο της ε, στρατηγικής μας. Και κάποια στιγμή ο κύριος Κάλλας, ο κύριος Μπαρόσο ε, ενδιαφέρονται σε σχέση με την ε, ακρόαση που ήδη προηγήθηκε στο Κοινοβούλιο. Οπότε θέλουμε και εμεί να δούμε πώ οι υποδομέ είναι πιο αποτελεσματικέ, όχι μόνο για τι οδικέ μεταφορέ, αλλά πάσα η υποδομή των μεταφορών. Άρα να δούμε πώ θα είναι πιο φιλικέ στο περιβάλλον μεταφορέ, πώ θα έχουμε κάποια οχήματα που μολύνουν λιγότερο. Όλα τα οχήματα. Και τα τρένα ακόμα. τελευταίο πάρα πολύ σημαντικό είναι το ότι πέραν πάσα συζητήσει όσον αφορά το πολιτικά το ζήτημα τη, της, κάποιων πόρων είναι γεγονός ότι η εσωτερήκευση τέτοιων δαπανών είναι κάτι το οποίο αφορά τους χρήστες και αυτό ε, σημαίνει ότι θα υπάρξουν ε, πλέον κεφάλαια για τις μεταφορές. Άρα έτσι ε, θα δούμε πώς θα μετακυληθούν αυτές οι δαπάνες και να, ε, δούμε, δούμε κατά πόσον ε, θα αποφύγουμε το να τιμωρήσουμε ε, τις οδικές μεταφορές ούτως υπήν ούτως ώστε να καταλήξουμε στην μετακίνηση των μεταφορών δια του σιδεροδρόμου. όχι θέλουμε ένα σύστημα το οποίο να έχει διαφάνεια να είναι δίκαιο ε, με τιμολογική πολιτική δίκαιη που να αντιστοιχεί στι ανάγκες των υποδομών. επομένως να δώσουμε αυτό το μήνυμα στου ε, operators και έτσι οι επιλογές του καθενός όσον αφορά τον τρόπο μεταφοράς να είναι τέτοιε επιλογέ οι οποίες να αντιστοιχούν όσο γίνεται πιο πιστά εις την γενική οικονομική λογική. Ε, να δούμε τώρα την επόμενη διαφάνεια. Είναι ευρύ αυτή η στρατηγική της εσωτερικής των δαπανών. Από το 2001 με κοινή τη Λευκή αρχίσαμε να συζητούμε για αυτή την κίνηση. Βεβαίω δεν και τίποτα γιγαντιαία το πρώτου, όμως το 2008 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέβασε αυτό, τη δέσμη ε, πράσινων μέτρων Ε, το 80% είναι η μεταφορά των εμπορευμάτων σε σχέση με το τι γίνεται όσον αφορά τις ε, χερσαίες μεταφορές. Και αντίστοιχο είναι και το ενδιαφέρον μας όσον αφορά την πολιτική αυτή τη οδηγήψη τη δαπάνη. Όμω λοιπόν να καλύψουμε ε, εν όχι μόνο τι σχετικέ μεταφορέ, αλλά όλου του είδου μεταφορέ, δηλαδή και, και του δρόμου και τι ενεργέ μεταφορέ και τι θαλασσίε, αλλά και την ιστορική ναυσιπλοεία. Οπότε όλα αυτά και τα περί των ανοιχτών ουρανών, όλα αυτά που σκοπούν στο να είμαστε πιο αποτελεσματικοί στι μεταφορέ, να καταναλώνουμε λιγότερη ενέργεια και επομένω να είναι κάτι το πιο βιώσιμο. Όσο αφορά τώρα του σιδηροδρόμου και τη σχετική νομοθεσία, μπορούμε εδώ πέρα να στοχεύσουμε αυτέ τι δαπάνε. Κυρίως μια που Προτάσει που θα κατεβάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εάν τελικά προωθηθεί η πρώτη δέσμη μέτρων για τους δρόμους, θα καλύψουν και αυτό το σημείο. Τέλος όσον αφορά τις θαλάσσιες μεταφορές. Έχει τοποθετηθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι εξορισμού είναι παγκόσμιο χαρακτήρα αυτές οι μεταφορές και επομένως πρόοδος θα σημειωθεί αν όχι από τον IMO θα γίνει τότε η πρόοδος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που θα κατεβάσει τις προτάσεις της. Έχουμε και κάποιες συνοδευτικά μέτρα αυτής της στρατηγική και κατά αυτόν τον τρόπο θα προωθήσουμε επενδύσεις για νέες τεχνολογίες, νέα πρότυπα όχι μόνο για τα οχήματα αλλά ακόμα και για τα διόδια. Πότε έχουμε διόδια στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οπότε θα είναι πάρα πολύ αναγκαίο να έχουμε κάποιο είδου διαλειτουργικά συστήματα πράξη των ε, διοδίων, ώστε να μην ε, διαταράσσουν, να μην ενοχλούνται οι οδικέ μεταφορέ. Το σταμάτημα, το φρενάρισμα, εκεί, στα, εκεί που καταβάζει στους σταθμούς διοδίων κλπ. Έχουμε μόνο σε ένα ευρωπαϊκό σύστημα διοδίων. Χρειάζεται κάτι τέτοιο και μέχρι το 2012 να έχουμε την αναγκαία νομοθεσία. Τότε να έχουμε δύο διαλειτουργικό σύστημα. Να είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί σε σχέση και με την ε, απόφαση για το ευρωπαϊκό αυτοκόλλητο σήμα την Ευρωβίνιατα. μόνο επομένως για μεταφορά εμπορευμάτων και βαρύ οχήματα σχετικά τώρα η Ευρωβινιέτα δεν αφορά άλλα οχήματα για τα επιβατικά, λεωφορεία είπαμε για τα διόδια που όπως έχει σήμερα η κατάσταση θα πρέπει να δούμε τη διαφοροποίηση σε σχέση με τόπο χρόνο και όχημα αλλά σήμερα μια που έχουμε τόσους περιορισμούς πρακτικούς για αυτή την ομοθεσία Πρέπει να κάνουμε κάτι γιατί δεν αποδίδει το σημερινό σύστημα. Δεν αποδίδει τόσο όσο θα θέλαμε να αποδίδει. Και για αυτό και θέλουμε να υπάρχει μια διαφοροποίηση πιο ξεκάθαρη όσον αφορά την, ε, την ε, πρότασή μας εδώ για την ε, Βροδινιέτα. Άλλωστε υπάρχει δέσμευση πολιτική μεταξύ Συμβουλίου και Οπότε αυτή η νέα πρόταση του ανάγκη 2006 ε, να μπορούμε να δούμε πώς δεν θα αντιστοιχεί στο κόστος της υποδομής όπως ισχύει σήμερα μπορεί να καλύπτει και άλλα εξωτερικά κόστη στο και δαπάνες. Αυτό αφορά πολλούς τρόπους μεταφορών. Και όπως σας προείπα, οι δύο τάξεις είναι ανεπαρκείς. Επομένως με τη νέα πρόταση θα μπορέσουμε να έχουμε εισπράξει και άλλων δαπανών θα μπορούσε κανείς να καλύψει διάφορα εξωτερικά κόστη Α δηλαδή, πούμε θα μπορούσε να, πεις, ε, να καλύψει το θόρυβο, την μόνιση του, της ατμοσφαίρας την προβολική κίνηση. Όμως τα κράτη-μέλη που θέλουν να θεσπίσουν τέτοιου είδους ε, τέλος θα πρέπει να υφετήσουν συγκεκριμένη μεθοδολογία και θα πρέπει τα έσοδα να χρησιμοποιηθούν για βιώσιμες μεταφορές. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό, μια που σήμερα η Γαλλία, το Βέλγιο, κάτω Σλοβακία και άλλα κράτη-μέλη έχουν εισαγάγει σιγά σιγά νέα συστήματα εισπραξής των 2-2. Ε, Όμως θα πρέπει να συμμορφωθούν προς την Ευρωβουλία και διαμορφώνει το ένα και αυτή η καινοτόμα τάση στα κράτη-μέλη. Νέοι τρόποι για να έχουμε διόδια τα οποία να αντιστοιχούν με το πραγματικό κόστος των μεταφόρων. Δεν έχουμε εναρμόνιση από πλευρά τη Ένωση. Όμω έτσι, ιδίω για τι περιφερειακέ χώρε, υπάρχει ο κίνδυνο να έχουμε συστήματα τα οποία διακρίνονται από δυσμενή, δυσμενείς διακρίσεις. Άρα η τα είναι μια εγγύηση για όλο τον κόσμο. και για τα κρατημέλη που είναι ας πούμε στο, πιο κοντά στο κέντρο της ε, Ένωσης αλλά και για τα πιο μακρινά, τα πιο περιφερειακά κράτη. Έτσι να έχουμε ένα σύστημα. Slide. Πάμε παρακάτω. Σας υπενθυμίζω πάντως ότι αυτό το που επιθυμούμε είναι να υποστηρίξουμε αυτή την πρόταση όχι μόνο με μια μελέτη επιπτώσεων όπως γίνεται συνήθως εδώ πως το πράγμα ήταν έτσι και πρωτότυπα μια που είχαμε εκατοντάδες σελίδων Είχαμε τεράστιες οικονομετρικές, οικονομικές μελέτες ε, για τα διαφορετικά μοντέλα. Όμως ε, έχουμε και μια επιπλέον μελέτη από το Κοινό Κέντρο Ερευνών, από αυτό το Ινστιτούτο της ε, Σεβίλης. Κατόπιν αιτήματος του Συμβουλίου ζητήσαμε να μας κάνουν μια μελέτη όσον αφορά τις επιπτώσεις για την μεταφορά την διασυνοριακή των προϊόντων τις στην τελική τιμή του προϊόντος και αυτό να, να, το κάνουν αφού λάβουν υπόψη την πρόταση της Κομισιόν μαζί με αυτά τα ανώρια, αυτά τα, ανώρια τα οποία εμείς εθεσπίσαμε με αυτή την πρότασή μας για να μπορέσουμε να αποφύγουμε υπερβολικές χρεώσεις πέραν των όσων θέλουμε απλώς οικονομικής και πολιτικής. Γιατί με αυτό το κοινό κέντρο ερευνών να κάνει μια τέτοια μελέτη και όχι μόνο για θεωρητικό μοντέλο αλλά να κάτσουν και να δούνε τι επιτόπου τι γίνεται να κάτσουν να πάρουν 5-6 διαδρομές διασυνοριακέ, να δούνε τι γίνεται σε σχέση με του κανόνες της πρότασή μα και να δουν να λάβουν υπόψη την, την, την, την ώρα εκκίνηση, την ώρα κατάληξη τι γίνεται όσον αφορά την κυκλοφορική συμφόρηση με τα συστήματα GPS οπότε για να δούμε τι γίνεται τώρα και γράψουμε παρακάτω την επόμενη διαφάνεια βλέπετε αυτό το, τον ε, διάδρομο Σινές Παρισίων έχουμε καμιά χιλιάδα προσωμιώσεις πάνω σε, αυτό το, σε αυτή τη διαδρομή. Με μεταβλητές, την ταχύτητα, τη λογική συμφόρηση κλπ. κλπ. Γιατί σας είπα δεν είναι εδώ πέρα θεωρητική αυτή η άσκηση πιχάρτου. Προσπαθούμε να δούμε οι καινούργιοι κανόνες τι επιπτώσεις έχουν στην πραγματική ζωή. Αυτή η διαδρομή Σινές Παρισιών είναι πάρα πολύ αντιπροσωπευτική περίπτωση διότι πρόκειται για ένα λιμάνι πάρα πολύ αναπτύσσεται ή στον Ατλαντικό, στην Πορτογαλία και το Παρίσι είναι ένα βασικό κέντρο από πλευρά οικονομία, από πλευρά δημογραφία. Είναι ένα εμπορικό, οικονομικό κέντρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε αυτή η διαδρομή είναι μια διαδρομή που πάρα πολύ συχνά ακολουθεί 144 χιλιόμετρα βλέπετε δεξιά σε αυτό το πλαίσιο τα αποτελέσματα δεν ξέρω αν είναι ευανάγνωστα βλέπετε ότι Ανα... όχι α έχετε πάρει κάποια αντίγραφα των διαφανειών Επόμενο, το κόστος είναι 2,9 ευρώ. Σεντ. Και ε, κυμαίνεται από 2,8 έως 3,4 δεκάρες αντίμ και το σύνολο είναι 54 ευρώ 2038 είναι το σύνολο οπότε περίπου έχουμε 2,5% ως αύξηση στο κόστος της μεταφοράς και σαν ε, ποσοστό της συνολικής επιβάρυνσης ε, έχουμε από όσον αφορά το θόρυβο 7% σύμφορες 6% και μόλι το 87% επομένω, βλέπετε εδώ πέρα ότι προκύπτει αβίαστα η εξήγηση ότι από την αρχή μέχρι το τέλος τη διαδρομής πληρώνεται η μόλις ατμόσφαιρα, από εκεί έχουμε τα διόδια ενώ η κυκλοφορική συμφόρηση πληρώνεται μόνο εκεί που υπάρχει συμφόρηση εκεί που είναι το κόκκινο και λιγότερο εκεί που είναι το πορτοκαλί στη διαδρομή. Τώρα, πάμε παρακάτω. Άλλο παράδειγμα. Τώρα, το, το, το, το χειρότερο σενάριο είναι αυτό το οποίο διαλέξαμε. Είναι επίση πάρα πολύ αντιπροσωπευτικό παράδειγμα, πάρα πολύ ρεαλιστικό. Σε πυκνοκατοικημένη περιοχή της Ευρώπης που έχουμε πάρα πολύ έντονη οικονομική δραστηριότητα, πολλέ μεταφορέ και αφορά εδώ πέρα κάποια βασικά οικονομικά κέντρα όπω η κολονία στη Γερμανία. Πιο μικρή αυτή εδώ με την προηγουμένη είναι 400-500 χιλιόμετρα. Εδώ όμω έχουμε πιο ακριβά διόδια. Το επιπλέον τέλος θα ήταν 5,3 cm ανά χιλιόμετρο. Και θα δοκιμαίνεται 4,2 ε, μέχρι τα 8,8 ως ε, ανώτατο ανά χιλιόμετρο. Και το σύνολο της επιβάρυνσης είναι το 5% του συνόλου του κόστου μεταφοράς και εδώ η κατανομή μεταξύ των επιμέρους χρεώσεων είναι 5% για το θόρυβο, 78% για τη μόνη ατμόσφαιρας και όμως εδώ έχουμε μεγαλύτερη χρέωση όσον αφορά την κυκλοφορική συμφόρηση που είναι 16%. Ζητήσαμε το Κοινό Κέντρο Ερευνών να υπολογίσει πώς αυτό θα επηρεάσει τις τιμές για τα προϊόντα τα οποία μεταφέρθηκαν με, τις, με τα μέσα αυτά. Πήραμε για παράδειγμα ένα μπισκότο, ένα, ένα φυλάτο τόνου, ε, ένα ζευγάρι jeans και ένα αυτοκίνητο. Και δώσανε μια τιμή ε, σε κάθε αντικείμενο. Ας πούμε τα τζιν είναι ακριβά τζιν, 50 ευρώ το πεντελόνι. Και το κόστος, η αύξηση του κόστους, όπως το διαβάζετε εδώ, είναι πάντα λιγότερο από το από 1%. Και για να μην πω και λιγότερο και από μισό της εκατό. Το μέγιστο της προσάυξησης είναι το φιλέτο τόνου που αυξάνεται κατά 0,34%. Τέλος πάντων, προσπαθώ να εισάγω και, μια, και λίγο χιούμορ σε αυτή την ε, συζήτηση. Αλλά τέλος πάντων, απλώς θα ήθελα να δείξω ποια είναι η συνεισφορά στην αύξηση του κόστους των προϊόντων που μεταφέρονται, που είναι αμεληταία θα έλεγα. Αυτό το οποίο δεν είναι... Το οποίο δεν είναι αμεληταίο, είναι το κόστος στους διαδρόμους αυτούς. Έχουμε έξι διαδρόμους και σας είχα δώσει κάποια παραδείγματα ε, δύο ε, διαδρόμων, Σινές Παρίσι και Ρότερνταμ ε, Κολονία. Λοιπόν, η... το... μέσο κόστος για τους έξι διαδρόμους είναι περίπου 4 σέντ ανά όχημα ανά χιλιόμετρο. Εάν υπολογίσετε, αν κάνετε όλους αυτούς τους υπολογισμούς σου, λαμβάνοντας υπόψη τα διόδια κτλ. κτλ έχουμε μια σημαντική αύξηση. κατά μέσον όρον η αύξηση του κόστους μεταφοράς είναι γύρω στο 3% και υπάρχει μια ε, διακύμανση των, ε, των αυξήσεων αυτών από 1,8 έως 5,2 στους διάφορους διαδρόμους. Τώρα, σύμφωνα με τα ε, υπάρχοντα διόδια που είναι 10 έως 30 σέντ ανά αυτοκίνητο ανά χιλιόμετρο θα υπάρξει μια αύξηση 25%. Και όπως σας είπα, επανερχόμενος και στην προηγούμενη διαφάνεια, όλες αυτές οι αυξήσεις, όλοι αυτοί οι υπολογισμοί δεν επηρεάζουν ε, σημαντικά την ε, τελική τιμή των προϊόντων. Επομένω, βλέπετε ότι και το κόστος δεν είναι, αν πείτε, θα μπορούσα να μου πείτε, και το, εφόσον το κόστος είναι, πολύ, είναι μεγάλο και ε, δεν επηρεάζονται οι τιμέ, γιατί τα κάνουμε όλα αυτά. Γιατί πιστεύουμε ότι ε, έχουμε μακροπρόθεσμα ωφέλη τα οποία ξεπερνούν κατά πολύ τα, ε, ε, τον αντίκτυπο των νέων διοδίδων, διοδίων. Συγγνώμη. Θα έχουμε βελτίωση στην αποτελεσματικότητα, θα έχουμε μακροπρόθεσμες ε, βελτιώσεις όσον αφορά την μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα, ε, την κυκλοφοριακή συμφόρηση θα έχουν, οι Ελβετοί έχουν κάνει συγκεκριμένες μελέτες και είδαν ότι παρόλο το ότι τα διόδια τους είναι πολύ υψηλά σε σχέση με τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά ε, όσον αφορά την, ε, τα φορτηγά είδαμε ότι οποιαδήποτε αύξηση που κάνουν είχε σαν αποτέλεσμα ένα, ε, μια πιο αποτελεσματική ε, κυκλοφορία των φορτηγών. Δεν υπήρχαν άδεια φορτηγά τα οποία να πηγαίνουν έρχονται. Και ούτως ή άλλως αυτό το οποίο θέλουμε είναι να ε, προσαρμοστούν και οι πρακτικές, αν θέλετε, ε, μετά την υιοθέτηση όλων αυτών των μέτρων. Τώρα, εάν λάβουμε υπόψη μας ε, την ε, κυκλοφοριακή συμφόρηση, θα έχουμε μία μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα λόγω ακριβώς της μειωμένης χρήσης των καυσίμων στις ε, οδικές μεταφορές. Και έγινε ο υπολογισμός και η μείωση αυτής της εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα θα ε, είναι περίπου 8% που δεν είναι αμεληταία μείωση. Και εάν ε, οι διάφοροι, διάφορες εταιρείες χρησιμοποιήσουν ε, με πιο ορθολογικό τρόπο την, τις μεταφορές, καλύτερες ώρες κτλ. Η μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης θα είναι 7% στους αυτοκινητοδρόμους και 10 με 30% στους τοπικούς δρόμους. Επίσης θα έχουμε κέρδη 2,3 ε, δισεκατομμύρια ευρώ ετήσια όσον αφορά την, ε, τις κοινωνικές δαπάνες και μέσω αυτού του συστήματος διοδίων, ε, αν χρησιμοποιηθεί σωστά δηλαδή το σύστημα, τα κράτη-μέλη θα έχουν ένα έσοδο που θα κυμαίνεται από 10-30 δισεκατομμύρια για την βιώσιμη κινητικότητα. Και δεν αναφερόμαστε εδώ, ε, δεν λαμβάνουμε υπόψη μας την, ε, το ότι θα πρέπει υποχρεωτικά οι πιστώσει αυτές και τα μέτρα αυτά να έχουν ε, συγκεκριμένο όνομα αν θέλετε. Τώρα, το εξωτερικό, οι, οι, χρεώ, χρεώσεις για το εξωτερικό κόστος θα αυξήσουν ε, κατά τη και μόνον το άμεσο κόστος των μεταφορών. Αυτό είναι ένα από τα συμπεράσματα στα οποία καταλήξαμε. Αλλά η αύξηση για τις ε, διεθνείς μεταφορές ε, με φορτηγά ε, θα είναι πολύ μικρή, πολύ περιορισμένη. Η... Αυτή που θέλουν να κάνουν τις μεταφορές ε, θα το οργανώσουν ε, πιο ορθολογικά, θα δούνε τι τους συμφέρει περισσότερο, ποια μέσα, μέσα μεταφοράς θα χρησιμοποιήσουν, ε, θα το δουν όλο αυτό με μεγαλύτερη προσοχή, θα το μελετήσουν. Η αύξηση του κόστους θα περιοριστεί εφόσον όλοι αυτοί θα προσαρμόσουν τις συμπεριφορές τους και θα αυξήσουν την αποτελεσματικότητά τους και το γενικό όμως όφελος της, ε, του υπολογισμού αυτού θα είναι πολύ σημαντικό. Θα έχουμε λιγότερη συμφόρηση, λιγότερες εκπομπές και παραπάνω χρήματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πασκούρα. Σας ευχαριστώ. Από το ΕΛΚ πρώτα. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Χαιρόμαστε που συζητάμε αυτή τη μελέτη σήμερα, ε, αλλά δεν συζητάμε ολόκληρη την έκθεση συνολικά. Αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει εμάς περισσότερο είναι αυτό το οποίο αναμένουμε εδώ και, δι... εδώ και μήνες. Την τοποθέτηση δηλαδή του Συμβουλίου. Γιατί βεβαίω είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η μελέτη, αλλά έχω την εντύπωση πως η μελέτη αυτή είχε στόχο να δώσει χρόνο στο Συμβούλιο να μην αποφασίσει και να μας πει εδώ πέρα κάτι το τελείως ασήμαντο για την Ευρωβινιέτα. Με τη μελέτη, εντάξει, ξέρουμε κάποια πράγματα παραπάνω, αλλά όχι εγώ προσωπικά, τουλάχιστον όχι πολύ περισσότερα. Δεν διάβασα ολόκληρη τη μελέτη, αλλά η εσωτερικοποίηση του κόστους, ε, κάτι το οποίο ήταν σημαντικό για εμάς ο ε, ΕΛΚΑ, ε, πρέπει να γίνει σε όλους τους τομείς, κάτι το οποίο εδώ πέρα δεν αναφέρεται, λέτε πως δεν ήταν στην εντολή σας. Και το ερώτημα μου είναι αυτό το οποίο αφορά βεβαίω ολόκληρο του ζητήματος του, της Ευρωβινιέτας. Τώρα για το κόστος της συμφόρησης, εγώ θα το έλεγα πλούστερα. Όποιος έχει το θάρρος να φορολογήσει μόνο τα φορτηγά ε, ενώ γνωρίζουμε πως δεν φταίνε μόνο τα φορτηγά για τη συμφόρηση αλλά και τα γεωταχή αλλά βεβαίως έχουν τελείως διαφορετικό λόμπι ίσως τότε νομίζω ότι δεν αντιμετωπίζουμε σωστά το πρόβλημα της συμφόρησης γιατί ήδη τιμωρείται ο επιχειρηματίας γιατί χάνει το χρόνο το φορτηγό του και πληρώνει τον οδηγό και αλλά από την άλλη πρέπει αν κάνει κανείς βόλτα ε, στο κέντρο του Στρασβούργου την ώρα που είναι κλειστά τα σχολεία ε, βλέπει πως δεν υπάρχουν εκεί πέρα μποτιλιαρίσματα εν πάση περιπτώσει όπως ε, σας είπα δεν προκαλούν μόνο τα φορτηγά συμφόρηση και εδώ πέρα απευθύνομαι και στην Κομισιόν. Σχεδόν καταφέρατε να δηλώσετε πως με την Ευρωβινιέτα δεν θα είναι πιο ακριβά τα πράγματα για τον επιχειρηματία, για τον καταναλωτή, αλλά θα προκύψουν πολλά λεφτά. Από πού θα έρθουν τα λεφτά. Γιατί λέτε πως πρέπει να οδηγηθούμε σε μια αλλαγή του μοντέλου η οποία θα προέλθει και από κάποιο κίνητρο το οποίο πρέπει να δημιουργηθεί για τον ένα ή τον άλλο τομέα. Οπότε ήταν φοβερή αυτή η αποστολή που είχατε, δηλαδή θα κοστίσει λίγο αφενός και από την άλλη πως τα λεφτά θα έχουν σημαντική επίδραση. Όπως σας είπα για μένα δεν έχει τόσο σημασία αυτό. Εγώ θέλω μία απάντηση στο απλό ερώτημα για τη δέσμευση των κονδυλίων. Τα λεφτά αυτά είναι απλά φορολογικά έσοδα ή θα προωθηθεί πραγματικότητα σε μία χώρα ή σε μία περιοχή. Και εδώ πέρα ούτε εδώ έρχεται αυτή η απάντηση γιατί είπατε πως πρέπει να βελτιωθεί η κινητικότητα χωρίς να διευκρινίσετε τίποτα άλλο. Γνωρίζω πως κάποιες χώρες ήδη με αυτό που ακούνε εκνευρίζονται. Ε, νομίζω το σημαντικότερο το οποίο μπορούμε να κάνουμε είναι αυτό, να απαντήσουμε αξιόπιστα σε αυτή την ερώτηση. Κατόπιν, εάν συγκρίνεται για τις ε, διαδρομές, ε, αναλύσατε είπατε δύο συγκεκριμένες διαδρομές αλλά ειλικρινά αν δούμε τη διαφορά ανάμεσα στο Euro 4 και στο Euro 5 σε μία από τις σημαντικότερες διαδρομές Rotterdam Κολονία και αν περάσουμε από το Euro 4 στο Euro 5 και ήμουν επιχειρηματία και έκανα μελέτη τι διαπίστωνα συνολικά ένα έπρεπε να αγοράσω ένα φορτηγό Euro 5 για να κερδίσω κάθε χρόνο 3.500 ευρώ. Παρά το ότι κάνω 300 διαδρομές ε, ετησίως ε, σε μία από τις πιο ακριβές διαδρομές. Δηλαδή τα νούμερα τα οποία μας δείχνετε εδώ πέρα δεν νομίζω ότι αποτελούν επαρκές κίνητρο για να αγοράσει κανείς ένα φορτηγό με προδιαγραφές Euro 5. δεν είναι και εδώ πέρα η συζήτηση αυτή των μέσων αλλά εν ολίγης, τα σημαντικότερα ερωτήματα δεν απαντήθηκαν και υπάρχουν α, ήδη από την αρχή της συζήτηση για την Ευρωβινιέτα. Όπως σας είπα ενδιαφέρουσα συζήτηση αλλά περισσότερο για το Συμβούλιο γιατί κερδίζει χρόνο και τρίτον ελπίζω η συζήτηση να γίνει πραγματικά με τη διαβούλευση με το Συμβούλιο και όχι με βάση θεωρητικές μελέτες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Γκρός. Εννέα ομιλητές έχουμε ακόμα. Γι' αυτό εδώ πέρα να υπενθυμίσω στους αδέλφους ότι θα είμαι αυστηρός. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πράγματι είναι φοβερά αυτά τα οποία λέει ο κύριος Γκρόση για την αιτία αυτής της μελέτης, ότι λέει θέλει να κερδίσει χρόνο το Συμβούλιο. Αλλά παρόλα αυτά νομίζω πως είναι απαραίτητο και για τους νέους συναδέλφους αλλά και για οποιονδήποτε παρακολουθεί αυτό τον φάκελο να δει λίγο σοβαρότερα τις συνέπειες εφαρμογής αυτής της οδηγίας. Και καλό είναι να ξεκινήσουμε υποθυμίζοντας πως αυτή τη στιγμή είναι απαγορευμένο να υπολογίσει κανείς το εξωτερικό κόστος και από ό,τι φαίνεται η εφαρμογή της οδηγίας ε, θα είναι κάτι το εθελοντικό, δεν είναι υποχρεωτική. Τέλο δεν θέλω να κάνουμε γενική συζήτηση, ας μείνουμε στη μελέτη. Τι βλέπω εδώ πέρα. Πρώτα απ' όλα, στην εφαρμογή των προτάσεων που υπάρχουν εδώ πέρα, πράγματι δεν υπολογίζονται όλα τα εξωτερικά κόστη και ειδικά από τα εξωτερικά κόστη τα οποία θέλουμε να ενσωματώσουμε, δεν υπολογίζεται ολόκληρη η πλήρη τιμή, αν θέλετε, για να διαπιστώσουμε κάτι. Δεύτερον, αντίκτυπος μειωμένο στο κόστος των μεταφορών, γύρω στο 3%, ένα 5,2% ως maximum υπολογίζεται. Τρίτον, σχεδόν καμία, κανένας αντίκτυπο στην τελική τιμή του προϊόντος για τον καταναλωτή. Επίσης διαπιστώνω πως παρόλα αυτά υπάρχει κάποιο αποτέλεσμα γιατί η μετάβαση από το Euro 4 στο Euro 5 θα έχει ένα ε, μπόνους, ένα όφελος όσον αφορά το κόστος, οπότε υπάρχει μια επιτάχυνση της ανανέωσης του στόλου και υπάρχει λοιπόν κάποια αύξηση της αποτελεσματικότητας και των πιο αηφόρων μέσων ε, μεταφοράς, αλλά για μένα σημαντικό είναι η διαπίστωση πως η οδηγία αυτή από μόνη της δεν επαρκεί για να οδηγηθούμε σε ένα πιο αηφόρο σύστημα μεταφορών είναι ένα μέσο μεταξύ άλλων, αλλά ένα σημαντικό στα μέτρα που θα πρέπει να λάβουμε τα επόμενα μέτρα για να επιτύχουμε τους στόχους μας. Είναι ουσιαστικό πράγματι να το επιτύχουμε αυτό. Κάτι άλλο το οποίο συμπεραίνω είναι πως ε, το κράτος θα πρέπει να αφιερώσει περισσότερα μέσα στην εφαρμογή και αυτό φαίνεται πως εάν και τα έσοδα τα οποία θα έχει χρησιμοποιηθούν καλά θα έχουμε ένα πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα δηλαδή θα μπορέσει να δώσει ακόμα περισσότερα πλέον εκτήματα τα οποία θα είναι μετρήσιμα αλλά τώρα το εάν θα δεσμευτούν για αυτή τη συγκεκριμένη χρήση τα, τα κονδύλια θα έχει πράγματι μεγάλο αποτέλεσμα στο εάν θα έχουμε τελικά θετική αξιολόγηση αυτής της οδηγίας. Επίσης αυτό το οποίο αναφέρεται για τη συμφόρηση. Χαίρομαι που ακούω πως ο Ματιέ είναι υπέρ του συμβιβασμού που είχα υποβάλλω, αλλά βεβαίως δεν το υποστήριξε η ομάδα του και λένε πως ε, στην περίπτωση που θέλουν τα κράτη-μέλη να κάνουν κάτι τέτοιο πρέπει να υπάρξει σύνδεση με άλλα οχήματα. Εδώ πέρα διαπιστώνω πως ε, η εφαρμογή αυτής της οδηγίας θα έχει ένα αποτελέσμα και θα είναι πολύ μεγαλύτερο πράγματι αν συμπεριληφθούν όχι μόνο τα φορτηγά αλλά και τα γιοταχή. Δύσκολη συζήτηση. Αλλά ας προσπαθήσουμε να βρούμε έναν ε, συμβιβασμό. Τέλος. Και ένα ερώτημα δηλαδή προς αυτούς που κάναν την μελέτη. Ποιο θα είναι το αποτέλεσμα στην περίπτωση στην οποία υπολογίσουμε πλήρως το κόστος της υποδομές. Καθώς εδώ πέρα μιλάτε μόνο για το εξωτερικό κόστος, ε, και θα μπορούσε να είναι πράγματι μεγαλύτερο στην περίπτωση που να και αυτό το οποίο ανέφερα. Εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι θετική ήταν αυτή η μελέτη και θα, μας, ε, θα αποτελέσει μια καλή εισαγωγή στην συζήτηση. Ευχαριστώ. Συνάδελφοι, είναι ενδιαφέρουσα η συζήτηση και πράγματι ανάβουν τα αίματα αλλά πρέπει να τελειώσουμε 6 ώρα για να ακολουθήσει και η συνεδρίαση των συντονιστών, οπότε σας παρακαλώ να είστε σύντομοι. Θα προσπαθήσω να δώσω τρία λεπτά σε όλους, ε, το οποίο βέβαια ξεπέρασε ο κύριος Αλχαντράου, η κυρία Πλασέρτ. Ευχαριστώ, θα είμαι σύντομη. Συγκεκριμένα ερωτήματα με τη μελέτη αυτή Ε, δεν ξέρω, ίσως απογοητεύομαι κάπως ε, καθώς ελπίζαμε πως θα έχουμε συγκεκριμένα μέτρα αλλά αν δούμε τις οδικές ε, μεταφορές βλέπουμε πως έχουν γίνει κάποια πράγματα τα προηγούμενα χρόνια και πλέον δεν υπάρχει περισσότερο περιθώριο για βελτίωση τη αποτελεσματικότητας από ό,τι αναφέρεται σε αυτή την έκθεση. Επίσης να αναφέρουμε τους χρόνους ε, φόρτωσης, εκφόρτωσης ε, και τα λοιπά. Επίσης, ε, νομίζω πως η χρέωση της συμφόρησης εδώ πέρα λάμβανε υπόψη πως συχνά δεν υπάρχουν άλλες εναλλακτικέ Αντιθέτως υποδεικνύει εδώ πέρα εναλλακτικές που δεν υπονοεί εναλλακτικές που δεν υπάρχουν. Και τέλος, θα μπορούσαμε αυτά τα ποσά να τα έχουμε σε ευρώ αντί για ποσοστά. Τέλος, όταν μιλάμε για 635 εκατομμύρια ευρώ είμαστε σε νούμερο του παρελθόντος. Ε, έχουμε φτάσει εντωμεταξύ στα 2,4 δις. Γιατί αυτή η διαφορά η οποία δεν είναι και πάρα πολύ καθησικαστική. Επίσης θα θέλαμε ακριβώς νούμερο ευρώ για το κόστος του συστήματος και το κοινωνικό κόστος και το κόστος της εταιρείας. συγκεκριμένα δηλαδή θέμε να ακούσουμε τα σωστά νούμερα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε λίγο. ο πρόεδρος Ναι, σας ευχαριστώ για την παρουσίαση της μελέτης. Συμφωνώ με τον συνάδελφο ότι δηλαδή εδώ πέρα το Συμβούλιο θα χαρεί για το ότι κερδίζει λίγο ακόμα χρόνο. Εάν όμως δούμε ακριβώς ε, τι μελέτη, υπάρχουν εδώ πέρα κάποια πράγματα τα οποία συζητάμε συνεχώς όπως ε, η επίδραση στις τελικές τιμές που δεν πρέπει να είναι πολύ υψηλή. Αναρωτιέμαι γιατί έγινε συζήτηση με το σύστημα ΙΑΣ που έχει υψηλότερες τιμές για να δούμε ποια είναι η ευελιξία του συστήματος. Νομίζω αυτό θα μας βοηθούσε πάρα πολύ περισσότερο και θα μας έδινε πολύ πιο ενδιαφέροντα αποτελέσματα για την περαιτέρω συζήτηση. Να υπενθυμίσω επίσης ε, κάτι άλλο. Είπατε πως ε, για να γίνει αποδεκτό θα πρέπει να υπάρξει οπωσδήποτε ένα όριο όσον αφορά τις τιμές και βεβαίως αυτό ισχύει πράγματι αν δούμε ειδικά το τι γίνεται με τους διαδρόμους αυτούς των ε, μεταφορών κοιτάξτε δεν ξέρω ε, είτε είναι μια τιμή η οποία είναι πολιτική τιμή είτε αλλιώς αναπτύσσουμε μαθηματικούς κανόνες ε, για το σύστημα και όχι κίνητρα. Δεν ξέρω, ίσως να μην διάβασα καλά επίσης Εγώ θα ήθελα κάποιες λεπτομέρειες ε, παραπάνω σε κάποια αισθήματα. Η αποτελεσματικότητα ενός μοντέλου, ειδικά όταν μιλάμε για τιμές, έχει ένα ανώτατο και ένα κατώτατο όριο. Θα ήταν δυνατόν να μου δώσετε τουλάχιστον ένα κατώτατο όριο αποτελεσματικότητας. Γιατί π.χ. αν δεν γίνεται τίποτα, δεν υπάρχει καμία αλλαγή κατά από τα 3-4 cents, δεν έχει κανένα νόημα να το εφαρμόσουν ε, και τα κράτη-μέλη. Γιατί δεν, δεν, δεν έχει μετά αποτέλεσμα. Οπότε η ελαστικότητα αυτού του μοντέλου προς τα κάτω θα έπρεπε λίγο να δοκιμαστεί. Αυτό το οποίο επίσης ε, με κάνει να απορώ είναι η εκτίμηση πως το σύστημα των διοδίων θα πρέπει να είναι συμβατό μέχρι το 2012. Δεν το βλέπω. Εάν δούμε τη συζήτηση καθώς έρχονται όλοι και λένε πως το δικό του σύστημα πρέπει να είναι το μοναδικό στην Ευρώπη και όχι τον άλλον, ε, δεν είμαι και πολύ αισιόδοξη. Δεν ξέρω πώς εσείς ε, φτάσατε σε αυτή την εκτίμηση. Δεύτερον, μιλήσατε για πιθανά μέτρα που θα αποτελούν διακριτική μεταχείριση στα κράτη, στην περιφέρεια της Ευρώπης. Να υπενθυμίσω πως αυτή τη στιγμή έχουμε μια κατάσταση που είναι διακριτική μεταχείριση όσον αφορά τα κράτη τα οποία είναι στο κέντρο και αποτελούν αν θέλετε κέντρο διερχομένων. Δηλαδή Ε, τα κράτη στην περιφέρεια της Ευρώπης είναι μόνο κράτη αφετηρίας ε, και προορισμού, ποτέ διερχομένων. Οπότε δεν ξέρω επίσης εάν ε, εδώ πέρα συμφωνεί με τους αρχικούς σκοπούς ο υπολογισμός συμφόρησης όπως τον έχετε κάνει. Ζέιλερ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Κοιτάξτε, υπάρχουν και κάποια νέα επιχειρήματα εδώ Παραδείγματο χάρη για την θέση που έχουν κρατήσει κάποια κράτη στο Συμβούλιο. Τα, το εξωτερικό κόστος λέγεται ότι έχει πληρωθεί ήδη, αλλά το πρόβλημα είναι ποιος το πληρώνει. Στην Λετωνία δεν έχουμε καν ούτε την πρώτη ευρωβινιέτ. Και ούτως ή άλλως πιστεύουμε ότι θα πρέπει να σκεφτούμε λίγο παραπάνω για την ε, νέα οδηγία για τα Ευρωβινιέτ. Π.χ. ας πούμε για την ατμοσφαιρική ρήπανση που και αυτή υπολογίζεται. Παραδείγματο χάρη στο συγκεκριμένο τομέα η απόφαση της Ρωσίας η οποία απαχορεύει από τους φορτηγατζίδες ε, από τη Λετωνία και την Λιθουανία να περάσουν τα σύνορα και που δημιουργούν, ε, δημιουργείται έτσι η μεγάλη συμφόρεση. Αυτό δεν είναι πρόβλημα της, ε, της Λετωνίας και μόνον, δεν ευθύνεται η Λετωνία γι' αυτό. Ε, επομένως βλέπετε κύριε Λίχτερμπερν ότι έχουμε, υπάρχουν πολλά προβλήματα. Και η έρευνα που έχει γίνει δείχνει ότι τελικά ούτω ή ο αντίκτυπος στην τελική τιμή του προϊόντων, των προϊόντων δεν είναι τόσο μεγάλος. Αλλά υπάρχουν και κάποιες χειροσκοπικέ κινήσεις. Και οι γεροσκοπικές κινήσεις που γίνονται στα καύσιμα ε, επηρεάζουν ούτως ή άλλως ε, την τελική τιμή και ίσως θα πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνουμε αποφάσεις. Θα ήθελα να πω όμως ότι εάν η χώρα σας πούμε δανειστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ούτως ή άλλως θα πρέπει να ξεχάσουμε τότε στην περίπτωση αυτή το κόστος αυτό, δηλαδή θα μπορούμε να το ε, υπολογίσουμε εσωτερικά πλέον. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος, όπως μας ζητήσατε. Πιστεύω ότι είναι ένα θέμα το οποίο το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ούτως ή άλλως δεν θα διαμορφώσουμε την άποψή μα ε, από τη μια στιγμή στην άλλη. Η πρόταση της Κομισιό μου θυμίζει το εξής. Ε, για να μην ε, δούμε την ασχήμια της, της νύφης ή του γαμπρού τέλος πάντων, μας παρουσιάζουν τον υποψήφιο ή την υποψήφια καλυμμένων. Τέλος πάντων. Το πρόβλημα είναι γιατί, γιατί γίνεται αυτή η πρόταση και δεν είναι ρητορικό το ερώτημα, η Κομισιό μας είπε ότι θα υπάρχουν, ε, θα υπάρχουν ε, μακροοικονομικά ε, συμφέροντα, τα οποία θα επικαλύπτουν κατά πολύ την, τις, τις δαπάνες και τα έξοδα που πρέπει να γίνουν. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι εδώ μιλάμε κυρίως για δικές μεταφορές και κυρίως μεταφορές μέσω των βαρέων οχημάτων. Χρειαζόμαστε χρόνο. Χρόνο για να εξετάσουμε όλα αυτά τα θέματα. Εγώ πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω πώς θα δεχτούμε την πρόταση αυτή, πώς μπορούμε να δεχτούμε την πρόταση αυτή. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι περνάμε μια οικονομική κρίση δεν μπορούμε να επιβαρύνουμε παραπάνω τις ε, μεταφορές. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι θαυμάσια αυτή η μελέτη της ε, Κομισιόν που δείχνει ένα πράγμα ξεκάθαρα. αυτοί που δεν πλήρωναν μέχρι τώρα για το κόστος τους δεν θα υποφέρουν. Κανείς δεν θα υποφέρει με την εισαγωγή αυτού του συστήματος. Εάν με είχατε πιστέψει δεν θα χρειαζόμασταν να κάνετε μελέτη, αλλά δεν με πιστεύατε. Εν πάση περιπτώσει. Προέκυψε αυτό το οποίο πάντα λέγαμε. Οι τιμές δεν θα ανέβουν. Επιτέλους θα εκπληρωθεί η αρχή ο πληρώνει αυτά τα οποία είχαν προβλέψει ότι θα βλαφτεί η οικονομία κτλ. δεν ισχύουν. Θα υπάρχουν πιο ήσυχα φορτηγά, πιο, με λιγότερο θόρυβο, λιγότερη συμφόρηση, μικρότερη κατανάλωση. Ωραία όλα αυτά. Ένα πράγμα δεν καταλαβαίνω. Από τη θέση της Κομισιόν. Όταν λέμε εδώ πέρα για μείωση του διοξιδίου του άνθρακα στις μεταφορές, όταν μιλάμε για προστασία του κλίματος, γιατί δεν συνυπολογίζετε τις εκπομπές και λέτε πως περιλαμβάνεται συμφόρηση. Λέτε πως είναι το 30% που είναι το υπόλοιπο 70%. Γιατί πνίγουμε τη βαριά βιομηχανία και θα φύγει τελείω από την Ευρώπη, αυτό θα γίνει, και δεν κάνετε εδώ πέρα τίποτα για τις μεταφορές. Δεν ξέρω. Θέλω μία απάντηση δεν είναι σαφές. Αν και εγώ ξέρω γιατί βεβαίως θα προέκυπτε πως δεν υπάρχει εδώ πέρα ούτε και με αυτό κανένα αρνητικό αποτέλεσμα. Νομίζω καιρό είναι να το σκεφτούμε. Μήπως δηλαδή ήταν λάθος ο δρόμος στον οποίο ακολουθήσαμε να μην συμπεριλάβουμε το διοξείδιο του άνθρακα. Ίσως έχω μια μικρή ελπίδα ότι μπορεί να μας βοηθήσει εδώ πέρα το Συμβούλιο με τις ε, καθυστερήσεις αυτές που έχει κάνει. Επιτέλους μπορεί τελικά να, να δράσει στο τέλος. Ευχαριστώ κυρία Φώστερ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σύντομη παρατήρηση θα ήθελα να κάνω. Δεν καταλαβαίνω τι γίνεται εδώ. Δεν καταλαβαίνω γιατί γίνονται, γιατί υπάρχει αυτή η έκθεση. Δεν νομίζω ότι μα βοηθάει και ιδιαίτερα έγινε πάρα πολύ δουλειά μεν, αλλά όλα αυτά τα ποσοστά 0,3, 0, κάτι, αυτά τα cents κτλ. κτλ σε, τι, σε τι ωφελούν όλα αυτά, μήπως μπορεί να είστε πιο συγκεκριμένοι. Έχουμε χάσει κάτι νομίζω. Πίσω στην τελευταία σελίδα λέει ότι εάν η, αν γίνουν δεκτές όλες αυτές ε, ε, οι προσαρμογές ε, θα, αυξηθεί, θα αυξηθούν τα, όχι μόνο οι οδικές μεταφορές αλλά και οι σιδηροδρομικές και θαλάσσιες κτλ. Μα το πρόβλημα ποιο είναι το ότι Το πρόβλημα είναι ότι ούτω ή άλλω υπάρχουν πιο πολλέ οδικέ μεταφορέ, διότι τα, οι είναι πιο ακριβη Και, σε, και σε σιδηρόδρομο πάλι να, να πα, εάν τυχόν πρέπει να γίνει συνδυασμό με θαλάσσιε μεταφορέ από το σταθμό μέχρι το πλοίο, τι θα γίνει. Πάλι οδικέ μεταφορέ θα χρησιμοποιήσουμε. Πάλι φορτηγά θα χρησιμοποιήσουμε. Λοιπόν, τώρα δεν ξέρω. Τα κράτη-μέλη θέλουν να εισάγουν διόδια, θέλουν να ε, κοστολογήσουν την ε, συμφόρεση, δεν ξέρω. Το πρόβλημα είναι και τα, πόσο, για πόσους τόνους μιλάμε, φορτικά πόσων τόνων μιλάμε. Τώρα το πρόβλημα δεν είναι τι λέμε εμείς, το πρόβλημα είναι και τι λένε και, η και τι λέει και όλος ο τομέας των βαρέων οχημάτων. Ο κύριος Κόκ. Ευχαριστώ κύριε Πασκαρέλη. Σέβομαι το έργο σας στην Κομισιόν Επίσης εξετάζω το αποτέλεσμα της μελέτης, αλλά έχω κάποιες αμφιβολίες. Πρώτα απ' όλα, εγώ θεωρώ πως υπάρχει εδώ πέρα πολύ μεγάλο γραφειοκρατικό έργο χωρίς συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Δεύτερον, τι μου δείχνει εμένα η μελέτη. Πρέπει να μιλήσουν επιτέλους οι μεταφορείς, γιατί δεν βλέπω εγώ κανένα κίνητρο να αγοράσουν καινούρια φορτηγά άμα περάσει αυτή η οδηγία. Και λέτε εδώ πέρα εάν ε, μειωθούν τα άδεια ταξίδια των φορτηγών. Πρέπει να δούμε τι θα γίνει και με το καμποτάζ. Νομίζω πως ε, δεν ξέρω ε, τι θα γίνει. Θα πρέπει να δούμε και τις οικολογικές διαδρομές. Και τέλος, και για να τελειώσω, συνεχώς νέα κονδύλια για την αϊφόρο μεταφορά όπω λέτε κτλ. Ε, το βρίσκω αστείο. Δίνονται εκεί πέρα περισσότερα λεφτά από όσα δίνει το γερμανικό κράτο αυτή τη στιγμή για την συντήρηση των δρόμων. Κύριε Φαντάλ, ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι ενδιαφέροντα τα αποτελέσματα της μελέτης. Μιλάτε για μία μικρή αύξηση 0,3 100 και για πολύ μικρό αρνητικό αποτέλεσμα το οποίο θα έχει. Δεν ξέρω αν θα το ερμηνεύα εγώ έτσι. Δεύτερον, τα συνολικά έσοδα, η κυρία Πλέσχορτ τα ανέφερε. Και εγώ έχω άλλα νούμερα, 2,4 δισεκατομμύρια και εγώ έχω πολύ χαμηλότερα νούμερα από αυτά. Και τέλος, εάν δούμε το συνολικό κόστος να αυξηθεί κατά 0,5% τι σημαίνει αυτό δηλαδή για την ε, Ολλανδία αυτό σημαίνει μια αύξηση 1 δισεκατομμύριο και σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση μεταξύ 10 και 15 δισεκατομμυρίων και εάν αποφέρει 12,4 δεν έχουμε κανένα αποτέλεσμα. Πρέπει δηλαδή να δούμε ποιο είναι το, η σχέση κόστους και ωφέλους. Απάντηση λοιπόν στο συγκεκριμένο ερώτημα. Σας παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Φαντάλεν. Κύριε Πασκαρέλη λοιπόν. Ακούστηκαν κάποιες ερωτήσεις, κάποιες υποψίες πως η μελέτη απλά μόνο το Συμβούλιο βολεύει. Έχετε λοιπόν τον λόγο για να απαντήσετε στις ανησυχίες των βουλευτών. Θα προσπαθήσω πράγματι, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ που μου δίνετε και τον λόγο. Δεν ξέρω εάν ε, θα ικανοποιήσω τους βουλευτές. Δεν θα απαντήσω εγώ στα ζητήματα πολιτικής γιατί δεν συζητάμε την Ευρωβινιέτα, μιλάμε για την μελέτη εδώ πέρα που έγινε με μια επιστημονική μέθοδο και με τα καλύτερα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας στο κοινό κέντρο ερευνών για να υπολογίσουμε τι αποτέλεσμα θα έχει η Ευρωβινιέτα όπως την προτείνει η Κομισιόν στην πραγματικό κόσμο. Οπότε θα περιοριστώ εγώ μόνο στα ερωτήματα που φορούν την ίδια τη μελέτη και όχι την πρόταση της Κομισιόν. Πρώτα απ' όλα, Η μελέτη είναι αυτό που είναι. Δεν καλύπτει αυτά τα οποία καλύφθηκαν από αρκετές παρεμβάσεις εδώ πέρα, δηλαδή η επιλογή του μέσου μεταφοράς, το σχετικό κόστος σιδηρόδρομου ή φορτηγού, την πολιτική που πρέπει να ακολουθήσει η Ένωση για την εσωτερικοποίηση του εξωτερικού κόστου σε σχέση με, τις, με τα υπόλοιπα μέσα μεταφορά, Είχα πει κάποια πράγματα στην εισαγωγή μου, δεν θέλω να τα επαναλάβω. Γνωρίζουμε πως με την Ευρωβινιέτα ασχολούμαστε με ένα κομμάτι ενός ευρύτερου προβλήματος, αλλά είναι σημαντικό κομμάτι. Όπως νομίζω θα παραδεχτούν όλοι. Η ευθύνη για την συμφόρηση ε, δεν θα μπω τώρα στο, στα χωράφια της πολιτικής. Γνωρίζω πράγματι πως δεν προκαλούν μόνο τα φορτηγά της συμφόρησης στους δρόμους. Αλλά τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας, που μας δίνει συνθήκη δηλαδή για την πολιτική μεταφορά, δεν μας επιτρέπουν να σχοληθούμε με τα ΙΟΤΑΧΗ. Αυτό μπορεί να το κάνω τα τη μελη Και οι τροπολογίες που πρότεινε ο κύριος Χαντραουή στην έκθεσή του πέρσι που την και το Συμβούλιο πηγαίνουν προς την ίδια κατεύθυνση. Δηλαδή αναγνωρίζουμε πως ε, οι αιτίες της συμφόρησης δεν είναι μόνο μία κατηγορία χρηστών. Πρέπει λοιπόν να έχουμε μία ολιστική προσέγγιση χρησιμοποιώντας και κοινωνικά και εθνικά μέσα. Η κυρία Χάνες Πλασκέτ ε, αν κατάλαβα καλά την παρέμβασή της, αναρωτήθηκε εάν οι διάφορες εξομοιώσεις ε, λαμβάνουν υπόψη τους κανονισμούς ε, περί ορών, οδήγησης, ε, ανάπαυσης κτλ. Και η απάντηση είναι ναι πράγματι. Επίσης ήθελε να γνωρίζει το κόστος Αυτό εξαρτάται από τις επιλογές που θα κάνουν τα κράτη-μέλη και την διαθεσιμότητα των ηλεκτρονικών διοδίων που είπε η κυρία Λίχτενμπέργκερ. Το εάν δηλαδή θα υπάρχει διαλειτουργικότητα το 2012. Ε, αυτό προβλέπεται. Δεν μιλάμε για εναρμόνιση, ένα ενιαίο σύστημα. Μιλάμε για διαλειτουργικότητα ανάλογα με τα συστήματα, δηλαδή τα διάφορα συστήματα που είναι να λειτουργούν μεταξύ τους. Και βεβαίω αυτό δεν αφορά μόνο τις μελέτες αλλά και τις δραστηριότητε όσων έχουν την, ε, το δικαίωμα χρήσης αυτοκινητοδρόμου που έχουν δεσμευτεί να γίνουν όλα αυτά μέχρι το 2012. Όπως σας είπα, το κόστος ε, εξαρτάται από την πραγματική κατάσταση, στην επιλογή των κρατών μελών και του τι υπάρχει ήδη. Δηλαδή το να στηθεί ένα σύστημα από το μηδέν σε ένα σύστημα διευρωπαϊκού δικτύου όπου αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν διόδια, οπωσδήποτε είναι πιο σοβαρό από το να προσθεθεί ένα κομματάκι σε ένα σύστημα που υπάρχει ήδη. Και εκεί που υπάρχει ήδη η τωρινή Ευρωβινιέτα, αλλά θα επανέλθω στην αξιολόγηση αντικτύπου που έχει ένα τμήμα για το κόστος ε, συναλλαγών του συστήματος. Δεν μπορώ τώρα να το συνοψίσω σύντομα. Τα 2,3 ε, δισεκατομμύρια ωφέλου στην κοινωνία στις μελέτες. Υπάρχουν εδώ πέρα κάποιες υποθέσεις που γίνονται και με βάση κάποιες υποθέσεις καταλήγουμε σε κάποια συμπεράσματα. και έχουμε εδώ πέρα τα ωφέλη ανακατηγορία υπολογίση, δεν θα τα επαναλάβω. Είναι όπως σας είπα μια πρόβλεψη που γίνεται με βάση κάποιες υποθέσεις και με βάση την εμπειρία. Αλλά έχουμε συνοψίσει τη, τη μείωση από την αλλαγή του μοντέλου, μείωση στον θόρυβο, φθορά υποδομών, κλιματική αλλαγή, ανανέωση στόλου, μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, μείωση της ατμοσφαιρικής ρήπανσης, μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα των οδικών μεταφορών. Ανέφερα πως η απάντηση των ε, εταιριών στις διαδοχικές αυξήσεις ε, των ελβετικών διοδίων ήταν αύξηση της αποτελεσματικότητας χρήσης των οχημάτων, δηλαδή δεν επέστρεφαν άδεια, είχαν περισσότερα φορτία κτλ. Και αυτό συνέβη και στη Γερμανία από όταν μπήκε το διόδιο εκεί για τα φορτηγά. Αυτά λοιπόν συνολικά. Μια αναφορά έγινε στην εξοικονόμηση εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Κύριε Λίχτρη, δεν είμαι σίγουρος ότι σας κατάλαβα. Αυτό το οποίο είπα. Για κάποιους λόγους που εξηγήσαμε και στην έκθεση του κυρίου Αλχαντραουή, η Κομισιόν έκανε μια πολιτική επιλογή να μην συμπεριλάβει το διοξείδιο του άνθρακα Αλλά εφόσον το διοξίδιο του άνθρακα εκπέμπεται στην ατμόσφαιρα με την καύση υδρογόνων ανθράκων, η μείωση της συμφόρησης με το τέλος συμφόρησης έχει συνυπολογιστεί στο τι αντιστοιχεί σε μείωση του διοξιδίου του άνθρακα. Γύρω στο 8% δηλαδή. Αυτά μπορώ να πω, αλλά βέβαιω πάντα η Κομισιόν είναι διαθέσιμη για περαιτέρω εξηγήσεις. Αν το επιθυμείτε κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τα μέλη. Τελειώνει εδώ πέρα η συνεδρίασή μας. Ε, ακολουθεί η συνεδρίαση των συντονιστών. Να υπενθυμίσω συναδέλφους πως ξανά αύριο στις 3 η ώρα το απόγευμα συνεδριάζουμε στην ίδια αίθουσα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τους διερμηνείς και στις ε, καμπίνες και τους ε, διερμηνείς